Good morning, ladies and gentlemen. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Θα αρχίσουμε. Γιατί έχουμε πολλά θέματα. Στις 10 πρέπει να αρχίσουμε την ψηφοφορία. 10 ακριβώς. Χρειαζόμαστε όλοι τις κάρτες μας για την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Εγώ ήδη τη βάζω στη θέση της. Λέξτε κι εσείς αν έχετε την κάρτα σας γιατί σε μία ώρα θα αρχίσουμε να ψηφίζουμε. Και είναι πολύ σημαντικό να έχετε την κάρτα σας στη θέση της για την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αρχίζουμε λοιπόν με το σημείο αριθμός 8. Είναι παρουσίαση της μελέτης πώς μπορεί η ευρωπαϊκή βιομηχανία να συμβάλλει στην ανάπτυξη και να ενισχύσει την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Επιτρέψτε μου να καλωσορίσω εδώ την κυρία Γιάννη Σέλβες που είναι από το Δανέζικο Τεχνολογικό Ινστιτούτο. Εσείς θα μας παρουσιάσετε το θέμα αυτό, σωστά. Κυρία μου, χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρίσκεστε εδώ μαζί μας σήμερα. Μετά θα ακούσουμε και παρατηρήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα προχωρήσουμε το θέμα και στην γραμματεία της Επιτροπής μας. Αλλά πρώτα απ' όλα να πούμε για αυτόν που έκανε τη μελέτη. Η μελέτη περιγράφει γνώσεις και προτείνει επιλογές προκειμένου η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία να συνεισφέρει στην αηφόρο ανάπτυξη. Πολύ σημαντικό θέμα για την Επιτροπή μας. Είναι πολύ σημαντικό να έρθουν επίσης τα εμπόδια και η παρουσίαση κάνει συστάσεις. συνθήκες, οι που πρέπει να ισχύουν για τις ε, εταιρείε μας κλπ. Εμείς ως πολιτικοί και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιστεύουμε ότι πρέπει να εξετάζουμε ξανά και ξανά αυτά τα θέματα ώστε να επανατοποθετούμεθα ανάλογα με τις συνθήκες. Είμαστε λοιπόν στο σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης. Έχετε το λόγο. Και καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ για την ευκαιρία αυτή που μου δίνετε. Είναι ένα μεγάλο θέμα το πώς δηλαδή η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία μπορεί να συνεισφέρει στην ανάπτυξη και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Δεν έχουμε την πλήρη απάντηση βέβαια, αλλά κάποια μηνύματα, κάποιες ιδέες θα σας τις μεταφέρουμε σήμερα. Πρώτα απ' όλα, όπως σίγουρα γνωρίζετε, η βιομηχανία είναι κλάδος κλειδί στην οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης. Είναι και υπηρεσίε βέβαια, αλλά και βιομηχανία μπορεί να συνεισφέρει στην οικονομική ανάκαμψη. Υπάρχει λοιπόν μια νέα αντίληψη για το ρόλο του κατασκευαστικού κλάδου στην διαδικασία αυτή που συνδέεται άμεσα με προστιθέμενη αξία, με γνώση και εντατικές υπηρεσίες. Στόχος της μελέτης αυτής είναι να σας ενημερώσουμε που βρίσκεται σήμερα η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία και πώς ε, μπορεί να τοποθετηθεί εκ νέου. Ποια είναι τα εμπόδια που αντιμετωπίζει η βιομηχανία αυτή, βέβαια υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες. Και συχνά οι παράγοντες είναι και εμπόδια αλλά και αδυναμίες που έχει ο ίδιος ο κλάδος. Συχνά υπάρχουν και τα δύο. Εμείς επικεντρωνόμαστε λοιπόν στις προποθέσεις εκείνες που μπορούμε να επηρεάσουμε και υπογραμμίζουμε το τι μπορεί να κάνει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση πολλοί βέβαια παράγοντες βρίσκονται εκτός ελέγχου των ευρωπαϊκών αρχών, αλλά παρόλα αυτά μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα για να αλλάξουν τα πλαίσια και να δημιουργηθούν οι καλύτερες δυνατόν προϋποθέσεις για την ενίσχυση της βιομηχανίας. Πρώτα απ' όλα λοιπόν να δούμε λιγάκι ποια είναι η κατάσταση πραγμάτων σήμερα. Γνωρίζετε δίχως άλλο ότι η ευρωπαϊκή ανάπτυξη δεν είναι όπως ήταν. Πριν από 14-15 χρόνια είχαμε την ίδια ανάπτυξη με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις χώρες του ΟΣΑ και μεγαλύτερη ανάπτυξη από ό,τι είχε η Ιαπωνία. Όμως η Ευρώπη δεν ανέκαμψε όπως άλλες περιοχές του κόσμου μετά την κρίση του 2008 και η ανάπτυξη φαίνεται ότι θα παραμείνει χαμηλή τα επόμενα χρόνια. Αν συγκρίνουμε την κατάσταση με τις Ομένες Πολιτείες όπου υπήρξε ανεργία, σταθεροποιήθηκε κάπως η κατάσταση το 2009, ενώ στη δικιά μας την περίπτωση έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα ανεργίας. Σήμερα στον κατασκευαστικό τομέα έχουμε 16% περισσότερο έχουμε μάλλον 16% ε, της συνολικής απασχόλησης, ενώ το 1995 ο κατασκευαστικός τομέας ήταν υπεύθυνος για το 21% της απασχόλησης. Από όλη θέσεων απασχόλησης επίσης ε, έχει επηρεαστεί πολύ και από, την, από τα χαμηλά προσόντα των εργαζόμενων. Τομείς ε, ψηλών τεχνολογιών έχουν ανακάμψει καλύτερα μετά την κρίση από ότι άλλοι τομείς που απαιτούν μεσαία ή και χαμηλού επίπεδου τεχνολογία. Ποιοι είναι λοιπόν οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα. Ο καθηγητής του Harvard, Michael Porter, είπε ότι όλα έχουν σημασία για την ανταγωνιστικότητα και μιλάμε εδώ πέρα για ανταγωνιστικότητα και σε ατομικές επιχειρήσεις και σε μεγάλους βιομηχανικού τομείς και στην εθνική αλλά και τη διεθνή οικονομία γενικότερα. Προσπαθούμε λοιπόν να ταξινομήσουμε τους παράγοντες αυτούς και εξετάζουμε συνεπώς το ανθρώπινο κεφάλαιο, το εργατικό δυναμικό δηλαδή, το κεφάλαιο, τα χρήματα που διατίθενται, κοιτάμε τις υποδομές, τον εξοπλισμό, κοιτάμε την καινοτομία, πιο συγκεκριμένα την τεχνολογική πρόοδο, κοιτάμε την παραγωγή και την ε, αλυσίδα, κοιτάμε τη δημιουργία, την ανάπτυξη, κοιτάμε τις πωλήσει και τέλος εξετάζουμε και το διοικητικό πλαίσιο, τις διοικητικές απαιτήσεις και τις ρυθμίσεις που ισχύουν για τις επιχειρήσεις. Αυτό είναι λοιπόν ένας κατάλογος παραγόντων που εξετάζουμε στη μελέτη αυτή. Πρώτον λοιπόν, ανθρώπινο κεφάλαιο, εκπαίδευση και προσόντα, δεξιοτεχνίες. Πολύ σημαντικό για να διατηρήσουμε και να αυξήσουμε την απασχόληση στη βιομηχανία. Το μήνυμα κλειδί, το ότι υπάρχουν διαφορετικές αλλαγές στο κατασκευαστικό τομέα, είναι κάτι που επηρεάζει πάρα πολύ και τις απαιτήσει για δεξιοτεχνίες στο εργατικό δυναμικό στο μέλλον. Όλο και περισσότερο βλέπουμε συστήματα προηγμένα, αυτοματισμό, ε, βλέπουμε ανάγκη για ψηφιακούς χειρισμούς, πράγματα αναγκαία για την ευρωπαϊκή βιομηχανία προκειμένου να ενισχυθεί παραγωγικότητα και να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, να χρησιμοποιούμε πιο αποτελεσματικά τους πόρους που διαθέτουμε. Αυτό βέβαια μπορεί να σημαίνει ότι θα χαθούν θέσεις απασχόλησης εξαιτία του αυτοματισμού και της ψηφιοποίησης, αλλά ε, μπορεί και να αλλάξει, γιατί μπορεί αυτό να συνδυαστεί με την διατήρηση και την αύξηση της απασχόλησης. Εξαρτάται από το τι είδους εργατικό δυναμικό έχουμε στη διάθεσή μας και πώς το χρησιμοποιούμε στη βιομηχανία. Σημαίνει επίσης, αν εξετάσουμε το εργατικό δυναμικό, ότι πρέπει να έχουμε αρκετούς μηχανικούς, αρκετούς επιστήμονες με υψηλά προσόντα, υψηλό επίπεδο εκπαίδευση, αλλά πρέπει συγχρόνως να επικεντρωθούμε και στο επίπεδο των πιο χαμηλό, δηλαδή στους εργάτες οι οποίοι και αυτοί πρέπει να έχουν τα κατάλληλα προσόντα, τις κατάλληλες δεξιοτεχνίες για τα νέα συστήματα που χρησιμοποιούν στην βιομηχανία. Πρέπει να ξέρουν πώς θα χειριστούν διάφορα μηχανήματα αλλά και την ψηφιακή τεχνολογία. Έχω κρυώσει και γι' αυτό κάθε τόσο δίχω. Συγγνώμη, λέω μιλήτρια. Αυτό σημαίνει ότι εμείς συστήνουμε πως σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να επικεντρωθούμε στην ανάπτυξη δεξιοτεχνιών κατάλληλων. Να δούμε τι δεξιοτεχνίες μας χρειάζονται στο μέλλον για αυτά τα νέα συστήματα που χρησιμοποιεί ο κατασκευαστικός κλάδος. Αυτό σημαίνει επίσης ότι πρέπει να υπάρχει διαβίου κατάρτιση. Είναι μια γνωστή έννοια αυτή επιτάχυνση εκπαίδευσης και κατάρτισης για εργαζόμενους που ήδη βρίσκονται στην αγορά εργασίας, αλλά πρέπει να αποκτήσουν νέα προσόντα. Και βέβαια χρειάζεται πάντα πολύ καλή ενημέρωση και πληροφόρηση για το τι δεξιοτεχνίες χρειάζονται, άρα πρέπει να ελέγχουμε πάρα πολύ καλά τη ζήτηση και την προσφορά όσον αφορά τις δεξιοτεχνίες που απαιτεί η αγορά εργασίας. Μήπως θέλετε ζεστό τσάι, ίσως θα μπορούσε να βοηθήσει αυτό. Ευχαριστώ. Ένα άλλο, ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι η πρόσβαση βέβαια σε χρηματοδότηση. Και εδώ η επίπτωση της οικονομικής κρίσης πριν από πέντε χρόνια είναι ε, πολύ ουσιώδης. Επηρεάζει πάρα πολύ τις δυνατότητες που έχουν οι επιχειρήσεις να έχουν δανειοδότηση. Η κατάσταση βέβαια είναι διαφορετική από χώρα σε χώρα. Άλλες χώρες υποφέρουν περισσότερο από έλλειψη τέτοιων οικονομικών πόρων, άλλες λιγότερο. Πάντως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παντού έχουν υποφέρει. Είναι επίσης ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και οι κλάδοι που έχουν πιο μεγάλο ρίζοδα χρηματοδότησης. Σε πολλές επιχειρήσεις δεν είναι γνωστό για πόσο χρόνο θα υπάρχει η δανειοδότηση και είναι πολύ δύσκολο να προγραμματιστούν και να προγραμματίσουν ε, την ε, έρευνα και την ε, ανάπτυξή τους. Πρέπει όμως αυτό να γίνεται και για τις παλιές επιχειρήσεις και για τις νέες που πρέπει να έχουν πάντα νέες ευκαιρίες. Και πάλι λοιπόν εδώ είναι πολύ βασικό εθνικές αρχές επίπεδο κρατών μελών να μπορούν να έχουν αξιόπιστες πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση των μικρομεσαίων τους επιχειρήσεων ώστε να προλάβουν τα προβλήματα. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης τα προγράμματα έρευνας και άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα να διασφαλίζουν ότι οι πληρωμές θα γίνονται γρήγορα και ότι οι μικρές κυρίως επιχειρήσεις δεν θα αντιμετωπίζουν προβλήματα για μήνες ή και χρόνια ακόμα χρηματοδότησης. Συστήνουμε επίσης να αναλυθούν και παρετέρω βήματα για επενδυτικά κεφάλαια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα είναι μακράς διάρκειας. Έρχομαι τώρα στις υποδομές. Φυσικά και οι ψηφιακές υποδομές με τα νέα προηγμένα συστήματα αποτελούν στοιχείο κλειδί για τις εξελίξεις και ξέρουμε ότι στην Ευρώπη έχουμε επικεντρωθεί πολύ σε αυτό. Χρειάζονται λοιπόν τέτοιες νέες τεχνολογίες για τις υποδομές σε πολλούς ε, τομείς και για τη διασύνδεση επιχειρήσεων μεταξύ τους. Ένα άλλο στοιχείο κλειδί είναι η ενέργεια. Εδώ δεν είναι η ίδια κατάσταση παντού στην Ευρώπη. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Το κόστος της ενέργειας, για παράδειγμα, είναι μια διαφορά. Άρα χρειάζεται εδώ πέρα μια πιο συνεκτική ευρωπαϊκή πολιτική όσον αφορά την ενέργεια. Αυτό θα έκανε τη διαφορά. Επιπλέον η Ευρώπη βρίσκεται υπό πίεση σε σχέση με ανταγωνιστές στο διεθνές επίπεδο για το κόστος της ενέργειας. Στην ε, Αμερική οι τιμές είναι μερικές φορές οι μισές από το κόστος που έχει να πληρώσει η Ευρώπη για την ενέργεια. Έπειτα υπάρχουν ε, βέβαια και επιταχυνόμενες ε, αλλαγές προς την κατεύθυνση των ευφυών δικτύων για να μπορούμε πιο αποτελεσματικά να ελέγχουμε την, ε, ενέργεια και τη χρήση της. Όσον αφορά τώρα τις πρώτες ύλες. Μερικές φορές δεν υπάρχουν αρκετές πρώτες ύλες στην Ευρώπη ή υπάρχουν ε, σε χώρες οι οποίες θέλουν να κρατήσουν ε, τους, ε, τις πρώτες αυτές ύλες για τους αυτούς τους, όπως κάνει η Κίνα. Άρα λοιπόν το θέμα της διαθεσιμότητας και το θέμα του κόστους των πρώτων υλών είναι πολύ βασικός παράγοντας για την Ευρώπη. Έπειτα το εμπόριο σε πρώτες ύλες πρέπει να μπει στην πρώτη γραμμή την ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ένας άλλος παράγοντας πέρα από το εμπόριο είναι να χρησιμοποιήσουμε και καλύτερα τις ύλες που ήδη διαθέτουμε ή που έχουμε ήδη χρησιμοποιήσει. Άρα να υπάρξει μια κυκλική οικονομία και να λάβουμε υπόψη μας και την ανακύκλωση των πρώτων υλών του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, για παράδειγμα, γιατί πολλές πρώτες ύλες υπάρχουν στον ηλεκτρονικό αυτόν εξοπλισμό και θα έπρεπε να μπορούμε να ανακτήσουμε τις ύλε αυτές από τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιούμε πια. Όσον αφορά τώρα την τεχνολογική πρόοδο και την καινοτομία. Η Ευρώπη βρίσκεται πίσω από τις ΗΠΑ στον τομέα της καινοτομίας. Δεν φτάνει η έρευνά μας στην αγορά. Κάνουμε έρευνα, αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είμαστε τόσο καλοί όσοι οι ανταγωνιστές μας και δεν καταφέρνουμε να βάλουμε στην αγορά και να χρησιμοποιήσουν οι επιχειρήσεις τα προϊόντα τα οποία απορρέουν από τη δικιά μας έρευνα. Εδώ λοιπόν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Αυτό βέβαια αντιμετωπίζεται κάπως με το νέο πρόγραμμα Horizon, αλλά πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα. Υπάρχουν επίσης μεγάλες ε, διαφορές στις ε, επιδόσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κάποιες χώρες που τα καταφέρουν καλύτερα ακόμα και από τις Ηνωμένε Πολιτείες. Άλλες πάλι βρίσκονται πολύ πίσω. Το χάσμα δηλαδή είναι μεγάλο και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν δίνονται αρκετές επενδύσεις στις έρευνες στον κατασκευαστικό τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τις Ηνωμένε Πολιτείες η έρευνα σε σχέση, οι δαπάνε μάλλον στην έρευνα σε σχέση με το ΕΠ αυξάνει μεν, αλλά με την κρίση εδώ υπήρξαν ε, προβλήματα και ίσως γι' αυτό πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη όθηση στις επενδύσει από τον ιδιωτικό τομέα στην έρευνα. Τι συστήνουμε λοιπόν από πλευράς του δημοσίου τομέα προτείνουμε να επικεντρωθούμε περισσότερο στις ε, ε, προμήθειες αγοράζοντας νέα τεχνολογία και να αναπτύσσουμε νέα τεχνολογία κυρίως για τομείς κλειδιά όπως είναι η υγεία, η δημόσια ασφάλεια, το περιβάλλον, η ενέργεια κλπ. Αλλά και εδώ αυτό το βρίσκουμε στο πρόγραμμα ορίζων, αλλά και μπορούν να γίνουν ακόμα περισσότερα. Επίσης, διδακτορικά θα έπρεπε να επικεντρωθούν περισσότερο στην έρευνα, αλλά να προωθήσουμε και τα διδακτορικά αυτά, ώστε να, γίνουν, να φτάσουν στην αγορά, στις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις δηλαδή να τα βλέπουν πιο ελκυστικά τα διδακτορικά αυτά. Τώρα η παραγωγή. Ε, δεν θα ξοδέψω πολύ χρόνο εδώ. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι προκειμένου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μεγαλώσουν πρέπει να προμηθεύουν μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να γίνουν πιο διεθνείς, για να υπάρξει καινοτομία σε αυτές. Χρειάζεται δηλαδή συνεργασία ανάμεσα σε μικρότερες και μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Βλέπουμε όμως πως κάποιοι τομείς, παρόλο που έχουν χαμηλή παραγωγικότητα και ψηλούς μισθούς, παρόλα αυτά τα καταφέρνουν γιατί έχουν σωστούς στόχους που είναι μεγάλες αγορές και χρησιμοποιούν και προηγμένες υπηρεσίες. Η επιχειρηματικότητα τώρα συνδέεται πολύ με το πώς εντάσσονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε μεγαλύτερες αλυσίδες. Ίσως θα έπρεπε να επικεντρώνονται περισσότερο σε επιχειρήσεις που ήδη υπάρχουν και που μπορούν έτσι να στηρίξουν οι πιο μεγάλες τις πιο μικρές και όχι ο καθένας να είναι από, μόνος του απομονωμένος. Για τις αγορές, η ενιαία αγορά φυσικά είναι ένα μεγάλο θέμα, έχει πετύχει πάρα πολλά. Παρ' όλα αυτά εξακολουθούν να υπάρχουν φραγμοί και σε μεγάλο βαθμό εξαρτώνται από τις χώρες μέλη και από το βαθμό στον οποίο έχουν εφαρμόσει τις ευρωπαϊκές διατάξεις σχετικά με την ενή αγορά και κατά πώς εφαρμόζουν και την αρχή της αμοιβές αναγνώρισης αγαθών, υπηρεσιών, προσόντων κλπ. Αυτό δεν γίνεται πάντα καλά από, από τα κράτη-μέλη ή από τους διάφορους τομείς. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, βλέπουμε ότι χρειάζεται ενίσχυση της νομοθεσίας, κυρίως της εφαρμογής των νόμων και των μηχανισμών που προβλέπονται. Για τις εξωτερικές αγορές και εκεί υπάρχει μεγάλος προστατευτισμός ακόμα. Και αυτό πρέπει να το συμπεριλάβουμε στις διαπραγματεύσεις. Είμαι στο τέλος, είμαι στο τέλος. Ε, διοικητικό και ρυθμιστικό πλαίσιο. Και εδώ το βασικό μήνυμα είναι ότι δεν είναι τόσο νέα ρύθμιση που χρειάζεται, περισσότερο χρειάζεται ενίσχυση της εφαρμογής των ρυθμίσεων που ήδη υπάρχουν και ισχύουν και να υπάρξει ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ψηφιακές ε, λύσεις για να μειωθεί το διοικητικό άχθος που έχουν επιχειρήσεις. Αυτά έχω να πω. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία μου, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση, αλλά πάντοτε το σημαντικότερο, τουλάχιστον στις δικέ μας συνεδριάσει, είναι να υπάρξει και συζήτηση. Θα δώσω πρώτα το λόγο στους συντονιστέ μας, συντονιστές μας στον καθένα. Ο κύριο Κάριν είναι ο πρώτος. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την σύντομη αυτή παρουσίαση. Θα διαβάσω εγώ σίγουρα και το έγγραφο πιο διεξοδικά. Γίνονται διάφορα ερωτήματα και ζητήματα. Θα ήθελα να στήσω τη συνολική σας άποψη για αυτά που αναφέρατε. Διαφορά μεταξύ της κατάστασης στην Ευρώπη και στη ΣΥΠΑ. Βλέπουμε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείες αναπτύσσονται, εμείς όχι, στην Ευρώπη συνολικά. Υπάρχει κάποια ιστέρηση και αυτό προβλέπουν οι αναλυτές και για το μέλλον. Η ερώτηση μου είναι ποια είναι η βασική διαφορά μεταξύ των οικονομιών των δύο αυτών περιοχών. Και εμείς οι νομοθέτες που πρέπει να εστιάσουμε για να μειώσουμε το χάσμα. Πολλά αναφέρατε. Παραδείγματο χάρη, το ενεργειακό, ενεργειακό κόστο μόνο του όμω δεν είναι το κλειδί για την ανταγωνιστικότητα. Η Ρωσία έχει χαμηλότερο ενεργειακό κόστο, αλλά είναι εντελώ ανανταγωνιστική, μη ανταγωνιστική, γιατί ε, δεν επενδύει πουθενά το κόστος και η πρόσβαση στο κεφάλαιο, το κόστος του κεφαλαίου. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα. Το εργασιακό κόστος, οι εργασιακές δομές, η μετακίνηση του εργατικού δυναμικού, η στάση των εργοδοτών. Αυτό δεν το αναφέρατε βέβαια. Οι δεξιότητες του εργατικού δυναμικού. Το αναφέρατε αυτό. Πρόσβαση στην αγορά. Πού οδηγούν όλα αυτά. Μήπως ε, το ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι μια ενιαία αγορά με ένα νόμισμα ε, κάνει τη διαφορά, εφόσον στην Ευρώπη δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είναι αυτή η άποψή σας ή βλέπετε άλλως τα πράγματα. Κόφορτ, από την ομάδα των Σοσιαλιστών Δημοκρατών. Ευχαριστώ. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εξαιρετική σας παρουσίαση. Νομίζω ότι τονίσατε κάποια σημαντικά σημεία. Όταν αναφέρατε στο σημείο 5 θα πρέπει να ενταχθούμε ακόμα πιο πολύ σε αυτή την αγορά, ε, σε αυτή την αλυσίδα μάλλον προσθέμενης αξίας για να έχουμε ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη. Θα ήθελα να επεκταθείτε λίγο αν ε, λαμβάνετε υπόψη τις θεωρίες του Μάικλ Πότερ. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα. Κάτι άλλο που είπατε και σχετίζεται με τα υψηλά ποσοστά ανεργία στην Ευρώπη ήταν η ανάγκη να έχουμε ένα πλαίσιο εξειδικευμένο για τις δεξιότητες, παραδείγματο χάρη, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση νέων αλλά και ενηλίκων με τη διαβίου να αποκτήσουν δεξιότητες που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν πολύ εύκολα σε εταιρείε και στην αγορά εργασία εν γέννη. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο αυτό και θα ήθελα να επεκταθείτε λίγο στο τι δυνατότητε περαιτέρω συνεργασία υπάρχουν, παραδείγματο χάρη, ε, επαγγελματική εκπαίδευση, διαβίου μάθηση, η εκπαίδευση στο πλαίσιο τη επιχείρηση. Γκρομπάτσικ από την ομάδα ECR. Θα μιλήσω στη γλώσσα μου κι εγώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κυρία μου για την παρουσίαση αυτή και για το γεγονός ότι μπορούμε να συζητήσουμε το θέμα αυτό σήμερα. Εστιάζουμε στον ανταγωνισμό μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα όμως νομίζω πρέπει να μας απασχολήσει και το ζήτημα της έρευνας, ε, της ανάλυσης του εσωτερικού ανταγωνισμού. Ποιος είναι ε, ο βιομηχανικός εσωτερικός ανταγωνισμός που προκύπτει άμεσα και από τις πολιτικές που εφαρμόζουμε εδώ στην Ευρώπη. Έχουμε τη γεωρική μας πολιτική, έχουμε την αλληλευτική μας πολιτική, την ενεργειακή πολιτική. Υπάρχει όμως έλλειψη άλλων πολιτικών. Έτσι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ορισμένα πολύ σημαντικά ζητήματα, ιδίως ε, στο πεδίο της οικονομίας. Έρχομαι στην ναυτιλιακή οικονομία, στη θαλάσσια οικονομία, για παράδειγμα. Έχει πάψει να υφίσταται εντελώ σε ορισμένα κράτη-μέλη αυτή η πολιτική. Και αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίω ε, στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, χάνεται εντελώ η βιομηχανική βάση που είτε μετατοπίζεται σε άλλα μέρη ή ευνοούνται άλλες περιοχές της Ένωσης. Υπάρχουν έντονε δε μεταναστευτικέ ροέ εξαιτία του γεγονότο αυτού, καθώ ο κόσμο αναζητεί δουλειέ, αναζητεί θέσει εργασία. Εξού και το ερώτημά μου. Έχετε ερευνήσει, μελετήσει αυτό το θέμα. Αν μπορώ να το χαρακτηρίσω βιομηχανική εκροή από ορισμένε περιοχέ τη Ένωση σε άλλε. Επίσης, η εξαφάνιση βαριάς βιομηχανίας από κάποιες ε, περιοχές και η μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων αυτών στην Κίνα ή άλλες χώρες. Ο πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριος Τέλτσκα τώρα έχει το λόγο. Εκ μέρους της ομάδας Άλντε. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Νομίζω ότι ένας άλλος βουλευτής ε, είναι αυτό ο οποίο θα μιλήσει εκ μέρου της Άλντε. Εγώ ήθελα το λόγο, μπορώ να μιλήσω αργότερα. Yeah. Ναι, εσείς, εσείς κυρία μου, παρακαλώ. Εκ μέρους της Άλντε. Όχι. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω για την εξαιρετική παρουσίαση. Θα ήθελα να σας υποβάλω δύο ερωτήματα. Το πρώτο αφορά και στη δικαιοπέψη της ΗΠΑ, όπως ε, και σε έκαναν αυτή τη σύγκριση, ε, θέλω και εγώ να αναφερθώ σε αυτή την σύγκριση για την ε, μετεγκατάσταση επιχειρήσεων από την Ασία προς την υπηρετική χώρα reshoring όπως λέγεται, όχι υπεράκτης πλέον δηλαδή, εξωχώριες εκμεταλλεύσεις. Πώς βλέπετε εσείς και τι κάνουμε και στο high-tech, clean-tech, υψηλή τεχνολογία, καθαρή τεχνολογία, έρευνα και ανάπτυξη εκεί. Επίσης, οι άνεργοι, ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν περισσότεροι άνεργοι είναι ότι δεν έχουν προσόντα για να ανταποκριθούν σε απαιτήσει ε, των νέων αυτών ε, θέσεων εργασία σε αυτέ τι βιομηχανίε. Τι μπορούμε να διδαχθούμε λοιπόν από τι ΗΠΑ ή άλλε χώρε που είναι πιο επιτυχημένε από εμά και πώ μπορούμε να διασυνδέσουμε καλύτερα την εκπαίδευση με τι νέε θέσει εργασία και τι μπορούν να κάνουν οι ίδιε οι βιομηχανίε. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Βανιού Βουίτσεν είναι το όνομά σα. Καλά το είπα, λέει ο πρόεδρο ή όχι. Πολύ κοντά ήσασταν. σα συγχαίρω, λέει ο ομιλήτρια. Ακούσαμε λοιπόν την άλλη, λέει ο πρόεδρο και τώρα η Γκούε, ο κύριο Ηλικιώτης. Όχι. ποιο θα μιλήσει. Α, η κυρία Έρνστ, παρακαλώ. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι συντονιστή, Μόλις μπήκε όμως ο συντονιστής μας, γι' αυτό θα μιλήσω εγώ. Έχω λοιπόν τις εξής ερωτήσεις. Και ε, όσον αφορά την ICT, την ε, ε, πολιτική πληροφορική, είπατε πάρα πολλά, μιλήσατε για τις υποδομές που πρέπει να εξελιχθούν. Νομίζω λοιπόν ότι στον τομέα αυτό υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε τι ακριβώς πρέπει να γίνει κατά την άποψή σας τα επόμενα χρόνια σε αυτόν τον θέμα. Αυτά για την πληροφορική. Το δεύτερο θέμα είναι το εξής, η αμοιβαία αναγνώριση αναγνώριση των ε, δεξιοτήτων διασυνοριακά. Γιατί είναι τόσο χρονοβόρα διαδικασία. Μα ποιο είναι τελικά το πρόβλημα. Το πρόβλημα βρίσκεται στα κρατημέλη. Γιατί δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Εγώ το έχω συζητήσει αυτό σε πάρα πολλές ε, περιφέρειες και περιοχές και βλέπω ότι εξακολουθεί δυστυχώς να εφίσταται το πρόβλημα. Το τρίτο που δεν αναφέρατε είναι οι διαφορές ε, στην παραγωγή και την παραγωγικότητα. Μιλάμε για ε, τεράστιες διαφορές μεταξύ πλούσιων και ε, φτωχών χωρών, μεταξύ ανεπτυγμένης και λιγότερο ανεπτυγμένης βιομηχανίας και υπάρχουν χώρες βεβαίως οι οποίες μαστίζονται από την κρίση, ας πούμε Ελλάδα και Κύπρος. Κατά την άποψή σας, Πώς μπορεί στις χώρες αυτές να προαχθεί ο βιομηχανικός τομέας, γιατί αυτές το έχουν απολύτως ανάγκη, όπως και φτωχέ χώρες, όπως είναι η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Ποια είναι λοιπόν η στρατηγική για τις χώρες αυτές, αφενός που μαστίζονται από την ε, κρίση και αφετέρου πολύ φτωχέ χώρες όπως είναι η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Ε, ο κύριος Μπορέλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κοιτάξτε, κατά την άποψή μου, η βιομηχανική ανάκαμψη δεν μπορεί να αγνοήσει το φορολογικό καθεστώς ε, στα κράτη-μέλη της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παραδείγματο χάνει στην Ιταλία. Υπάρχει κάποια παραγωγικότητα, αλλά δεν μπορούν να επιτύχουν μεγαλύτερη πρόοδο οι ενδιαφερόμενες ε, επιχειρήσεις, γιατί υπάρχει δυστυχώς στραγγαλισμό σε φορολογικό επίπεδο. Και αυτό δεν νομίζω ότι ισχύει μόνο στην Ιταλία. Εγώ λοιπόν εύχομαι σύντομα να αρχίσει κανείς να σκέπτεται πώς είναι δυνατόν να μειωθεί η φορολογική πίεση στα κράτη-μέλη για να επιτευχθεί η ολοκλήρωση της κοινή αγοράς όπου όλοι θα ξεκινούν από την ίδια βάση. Επενδύσεις ε, πρέπει να γίνουν στην έρευνα και την τεχνολογία. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, βέβαια έχουν πολλές ε, δυσκολίες στο να ακολουθήσουν αυτή την εξέλιξη. Οι περισσότερες αγωνίζονται να επιβιώσουν σε μια αγορά η οποία είναι όλο και πιο ανταγωνιστική. Νομίζω λοιπόν ότι είναι απαραίτητη απαραίτητο να εργαστούμε όχι μόνο για την πρόσβαση στην πίστη, όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε, αλλά και στην κατάργηση των φόρων σε τέτοιου είδους επενδύσεις, έτσι ώστε να είναι πολύ πιο εύκολη η πρόσβαση σε αυτούς τους πόρους, να περιοριστεί και η γραφειοκρατία. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω ότι εγώ είμαι επιχειρηματίας ε, και δεν έχω ακούσει ποτέ να γίνεται λόγος για Enterprise Europe ε, Roadmap, και αυτό το άκουσα πρώτη φορά όταν έγινα Ευρωβουλευτής. Τον διακόπτη πρόεδρος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα λοιπόν, αν έχετε την καλοσύνη, να σχολιάσετε και να απαντήσετε στις ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω. Αν είχα απαντήσει όλα αυτά τα ερωτήματα, δεν θα καθόμουν μάλλον εδώ. Θα είχα πολύ ψηλότερη θέση. Θα κάνω πάντως ό,τι μπορώ. Λοιπόν, αρχικά, είχαμε ένα ερώτημα για τις διαφορές μεταξύ ΙΠΑ και Ευρωπαϊκής, μάλλον και Ευρώπης. Και ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες που εξηγούν αυτή την ε, καθυστέρηση. Εσείς αναφέρατε πολλούς από αυτούς τους παράγοντες. Δεν υπάρχει μία και μόνη εξήγηση. Νομίζω ότι το κόστος κεφαλαίου και η διαθεσιμότητα κεφαλαίου είναι ένα τεράστιο ζήτημα. τελευταία ήταν πιο εύκολο, ιδίως για το επιχειρηματικό κεφάλαιο ε, στις ε, Ηνωμένε Πολιτείες, ε, ενώ ήταν πάντα ένα μεγάλο ζήτημα για την Ευρώπη λόγω της τόσο μικρής διαθεσιμότητας σε σχέση με τη ΣΥΠΑ. Και κατά την άποψή μου, και εξ όσων γνωρίζω, είναι πολύ χειρότερο σήμερα το πρόβλημα. Το επιχειρηματικό κεφάλαιο έχει μειωθεί δραστικά. Κάτι άλλο που παρατηρούμε είναι ότι ενώ το δημόσιο μερίδιο του επιχειρηματικού κεφαλαίου μπορεί να ήταν 10-20% έχει ανέβει τώρα και ανέχεται περίπου στο ίμιση, ενώ το ιδιωτικό επιχειρηματικό κεφάλαιο έχει μειωθεί, έχει αντικατασταθεί από δημόσιο σε μεγάλο βαθμό. Αυτό λοιπόν είναι μια λύση, αλλά το ζήτημα είναι θέλουμε να συνεχιστεί αυτή η εξέλιξη. Δεν είμαι η Δήμων ε, σε ό,τι αφορά τι χρηματοπιστωτικές αγορέ, αλλά σίγουρα εσείς ε, οι ρυθμιστές, οι νομοθέτες πρέπει να εξετάσετε αυτό το ζήτημα του κόσμου του κεφαλού. Φόροι. Υπήρχαν πολλά ερωτήματα. Φυσικά και υπάρχουν φορολογικές διαφορές, είναι διαφορετικά τα φορολογικά καθεστώτα. Ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προνόμιο των κρατών μελών να καταρτίζουν τη φορολογική πολιτική. Γι' αυτό και δεν ε, πραγματευόμαστε αυτό το θέμα στην έκθεσή μας. Αν θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση κατόπιν προτάσεις του Κοινοβουλίου να ασχοληθεί με αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Προς το παρόν είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών να λάβουν τι αποφάσει. Και βέβαια το ζήτημα τη ενιαία αγορά. Είναι πολύ σημαντικό το αναφέρετε και εσεί οι ίδιοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια μεγάλη ενιαία αγορά που όμω έχει ακόμη πολύ σοβαρά προβλήματα. ίσως αυτό το ζήτημα είναι το πιο σημαντικό και πρέπει τα εμπόδια στην ενιαία αγορά να αντιμετωπιστούν από πλευρά των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Ο κ. Σκόφερ μίλησε για την παγκόσμια λυσίδα αξίας, την ανάγκη για δεξιότητες, για το πλαίσιο δεξιοτήτων. Ήδη έχουν αναλυφθεί αρκετές πρωτοβουλίες. Δεν θα σας τις αναφέρω. Πιστεύω όμως ότι πρώτα απ' όλα Υπάρχει ανάγκη να δίνεται καλύτερη ενημέρωση για τις ανάγκες σε ό,τι αφορά δεξιότητες. Και στατιστική μπορεί να βοηθήσει και υπεραιτέρω έρευνα μπορεί να βοηθήσει. ώστε να ρωτήσουμε τις ίδιες επιχειρήσεις τι χρειάζονται, ποιες δεξιότητες χρειάζονται. Και βέβαια εδώ υπάρχει ένα τεράστιο δυναμικό συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών. Ήδη βλέπουμε κάποιες πρωτοβουλίες Στη χημική βιομηχανία, για παράδειγμα, εξετάζεται αυτό το πλαίσιο δεξιοτήτων και ποια είναι, ποιες είναι οι ανάγκες. Θα μπορούσε λοιπόν να μιμηθούν και άλλες ε, βιομηχανίες το παράδειγμα αυτό. Ένα άλλο ερώτημα ήταν το κύριο Κοβάλτσο και κάπως έτσι, λυπούμε αν δεν προφέρω σωστά το όνομά σας. Το βασικό νομίζω ήταν οι διαρθρωτικές αλλαγές στη βιομηχανία, ιδίω στις ανατολικοευρωπαϊκές χώρες που έχουμε μεγάλο βαθμό από βιομηχάνηση που παρατηρείται αυτή η μετεγκατάσταση επιχειρήσεων και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες αλλά και εκτός Ευρώπης, σε άλλες περιοχές του κόσμου με χαμηλό κόστος εργασιακό. Ένα πολύ καλό παράδειγμα νομίζω είναι η Σλοβακία που έχει καταφέρει να ενσωματωθεί στις ε, ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας ιδίω στο τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Υπάρχουν διαφορές ακόμη ε, στο μισθολογικό και άλλο κόστος. Η Σλοβακία λοιπόν έχει προσελκύσει ξένες επενδύσεις, ιδίως από τη Γερμανία, όπου ε, έχει ανοίξει νέα εργοστάσια στη χώρα αυτή. Άρα δεν μιλάμε για μια νέα ροή εκτός Ευρώπης, υπάρχουν και εξέλιξεις εντός Ευρώπης για την αποβιομηχάνηση στην Ανατολική Ευρώπη δεν έχω λύσεις. Αλλά μπορείτε να διαβάσετε για μεγαλύτερες λεπτομέρειες το σχετικό κομμάτι της εκθεσής μας. Ρωτήσατε για το reshoring, της δεξιότητες. Αυτό το θέμα είναι τεράστιο. Δεν είμαι ειδική βέβαια. Βλέπουμε να υπάρχει μια αισθητή τάση. Επειδή υπάρχει ψηλό κόστος στην Κίνα πλέον και επειδή υπάρχει αυτή η εξάπλωση των αλυσίδων αξίας και το θέμα του ελέγχου ποιότητας, πόσα λεπτά έχω εσύ μου, λίγα, ε? Βλέπουμε λοιπόν μία με την κατάσταση επιχειρήσεων ε, όχι πλέον να έχουμε την αντίστροφη πορεία, reshoring και όχι ε, out offshoring μάλλον, έχουν γίνει πολλά για να οριστούν ε, οι ανάγκες σε δεξιότητες και αυτό είναι το πρώτο βήμα γιατί πρέπει να έχουμε το σωστό εργατικό δυναμικό με τις σωστές δεξιότητες. Έτσι θα παραμείνουν στην Ευρώπη οι βιομηχανίες. Για την αμοιβή αναγνώριση υπήρξε ένα ερώτημα Θα μπορούσαν οι ευρωπαϊκές, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να ασκήσουν κάποιες πιέσεις, αλλά τα κράτη-μέλη είναι αυτά που θα πρέπει να κάνουν τα βήματα ε, της αμοιβές αναγνώρισης ε, στα προσόντα, αλλά και σε αγαθά και υπηρεσίες σε διάφορα τομείς, γιατί αυτό είναι ένα τεράστιο εμπόδιο στην εσωτερική αγορά. Ναι, μεν υπάρχει ο, ο κανονισμός, υπάρχουν οι ρυθμίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν εφαρμόζονται πλήρως όμως από τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν πολλά εμπόδια. κ. Μπορέλη μίλησε για τους φόρους. Επαναλαμβάνω, είναι θέμα εθνικό, εθνική αρμοδιότητα. Αν το Κοινοβούλιο θέλει να ασχοληθεί, σίγουρα θα πρέπει να γίνουν ε, τεράστιες αλλαγές. Είναι γεγονός όμως ότι υπάρχει μεγάλη ε, διαφορά μεταξύ των φορολογικών συστημάτων και ανάλογα με το κράτος μέλος, κάποιες, ε, μάλλον οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν πολύ μεγάλο φόρτο, άλλες λιγότερο πρέπει να πληρώνουν διάφορες διοικητικές απαιτήσει. Σε κάποιες χώρες οι ΜΜΕ να τα βρίσκουν δύσκολα, σε άλλες όχι τόσο. Το ευρωπαϊκό πιο ένα τεράστιο δίκτυο αυτό. Πολλά μέλη του δικτύου είναι τοπικά εμπορικά επιμελητήρια. Θα μπορούσε να υπάρξει μια ευρύτερη διαδικασία ευαισθητοποίηση για να προσεγγίσουμε και άλλου επιχειρηματίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περνάμε τώρα στον επόμενο γύρο των ερωτήσεων. Θέλετε να διαμαρτυρηθείτε? Κοιτάξτε, μία ερώτηση δεν μου απαντήσατε, που είναι όμως πάρα πολύ σημαντική. Σας ε, ερώτησα για την βιομηχανία που αφορά χώρες που μαστίζονται από την κρίση, όπως Ελλάδα και Κύπρος ε, και άλλες φτωχές χώρες. Δεν είπατε τίποτα απολύτως, ανεξάρτητα από τη μελέτη σας, όμως εφόσον μιλάμε για την εκβιομηχάνηση στην Ευρώπη, νομίζω ότι αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, κοιτάξτε, θα σας απαντήσει η ομιλήτριά μας στο δεύτερο γύρο απαντήσεων, αν μου επιτρέπετε. Τώρα, έχουν ζητήσει το λόγο 10 ε, ευρωβουλευτές Άρα δηλαδή σας παρακαλώ να κάνετε ερωτήσεις ένα λεπτό ο καθένας ε, και αν έχει την να μην κάνετε τοποθετήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Η εικόνα που ε, σκιαγραφείτε δεν είναι καλή ε, τουλάχιστον όμως ε, αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα. Ε, το θέμα που θέλω να δείξω έχει σχέση με την εκπαίδευση, την έλλειψη εκπαιδευμένων μηχανικών ανθρώπων με διατριβή και ερωτώ αυτό το αντιμετωπίζετε και αν ναι πού. Γιατί αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το ελέγχουμε εμείς στην Ευρώπη και δεν νομίζω ότι πρέπει αυτό να δημιουργεί πρόβλημα. Πολύ ωραία λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Ντεκαστήλο Ντεκαστήλο η επόμενη μιλήτρια. Ευχαριστώ. Δεν έχω πολύ χρόνο βέβαια για να παρέμβω, αλλά γι' αυτό θα διαλέξω μόνο το θέμα της πρόσβασης στις αγορές. Αναφερθήκατε στην εσωτερική αγορά, που είναι και το στοιχείο κλειδί για την επαναβιομηχανοποίηση και για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Εδώ όμως το πρόβλημα είναι διτό. Το ένα είναι ότι υπάρχουν ναι, πολλά διοικητικά προβλήματα. Το ένα τρίτο ή τα τρίτο ή τα μισά διοικητικά προβλήματα που έχει η ευρωπαϊκή βιομηχανία έχει να κάνει με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και με θέματα εφαρμογής σε εθνικό επίπεδο. Αλλά το άλλο πρόβλημα είναι υπερβολικός κατακαιρματισμός στην νομοθεσία. Εδώ αναφέρεται ότι πρέπει να ενισχύσουμε την καλή εφαρμογή πολύ περισσότερο από όταν να φτιάξουμε νέα νομοθεσία. Εγώ νομίζω ότι χρειάζονται και τα δύο διότι για τα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει τεράστιο κατακαιρματισμό και ίσως και γι' αυτό να είναι πρόβλημα γιατί υπάρχει τεράστιος κατακαιρματισμός στη ρύθμιση στην Ευρώπη. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να σταθμίσουμε καλά τι έχουμε παραπάνω πόσο χρειαζόμαστε και τι δεν έχουμε αρκετά. Ευχαριστούμε. Τελίσκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για την εισήγηση που ακούσαμε. Κοιτάξτε, με εκπλήσει λιγάκι το γεγονός ότι δεν ακούσαμε να πείτε τίποτα για την βελτίωση των ε, ρυθμίσεων και κανονισμών. Πρέπει λοιπόν να είμαστε ειλικρινεί και να πούμε ότι ε, δεν είναι ότι εμείς ε, προσφέρουμε πάντα σωστούς κανονισμούς για να επιτύχουμε τους στόχους μας η Κομισιόν δεν ανταποκρίνεται, ούτε και το Συμβούλιο προβαίνει σε αξιολόγηση επιπτώσεων. Ίσως και το Κοινοβούλιο θα έπρεπε να τα καταφέρνει καλύτερα. Αυτό που είπατε για την επιχειρηματικότητα, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και θα πρέπει ίσως να το παρακολουθήσουμε, γιατί από ό,τι φαίνεται οι επιχειρηματίες μας δεν έχουν την δυνατότητα να ε, προοδεύσουν περισσότερο. Και κάτι άλλο. Υπάρχει και εσωτερικός προστατευτισμός. Στη τελική ανάλυση θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε καλύτερα ε, στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η εσωτερική αγορά. Ε, ναι, μεν ε, καταργούμε κάποιους φραγμούς, αλλά υπάρχουν ακόμα αρκετά συστημικά εμπόδια. Ο κύριος Ρόιλ, παρακαλώ. Καταρχήν θέλω να πω ότι η συζήτηση αυτή δείχνει ότι στην Ευρώπη πρέπει να συζητάμε επί της ουσίας περισσότερο, γιατί μέχρι τώρα ήμασταν πολύ επιφανειακοί. Αυτό ήταν το πρώτο το δεύτερο που θέλω να πω. Πρέπει η συγγήτρια να μας ενημερώσει καλύτερα για το ενεργειακό κόστος. Αυτό είναι ένας παράγον της βιομηχανίας. Και ποιες είναι οι συνέπειες. Πρέπει δηλαδή στην Ευρώπη να ασχοληθούμε με, την, με το fracking, με τη ρογμάτωση. Ε, θα πρέπει ίσως να ασχοληθούμε περισσότερο με τις ανώσιμες πηγές ενέργειας. Και το τρίτο ερώτημα είναι πώς μπορούμε να βρούμε κάποια λύση όταν λέτε η ίδια ότι πολλές φορές οι κανονισμοί είναι πολύ περίπλοκοι. Και αυτό ε, το βρίσκεται ενδιαφέρον. Κανεί δεν το έχει θίξει. Τι να κάνουμε, λιγότερους ε, κανόνες, λιγότερους νόμους ε, και να κοιτάμε έτσι ώστε να εφαρμόζονται οι παλιοί. Κατά την άποψή μου αυτό πρέπει να συμβεί. Αν όμως συμφωνούν όλοι, τότε αυτό θα πρέπει να έχει συνέπειε. Δηλαδή θα σημαίνει ότι στο μέλλον θα υπάρξει περιορισμός του νομοθετικού έργου. Θα ήθελα να επισημάνω, λέει ο κύριος Χένκελ, ότι δεν είναι χρήσιμο μόνο να συγκρινόμαστε με άλλους, αλλά να συγκρινόμαστε και με άλλους μέσα στην Ευρωζώνη. Για μένα είναι σαφές ότι η αποβιομηχάνηση γίνεται στο νότο της Ευρώπης και όχι στη δική μου τη χώρα. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω κατά πόσον συμφωνείτε με τη Βρετανική κυβέρνηση που λέει ότι το ευρώ είναι ας πούμε πολύ ισχυρό για τη Γαλλία, ίσως και για την Ιταλία και για άλλες χώρες ε, του Νότου και πολύ αδύναμο για τη Γερμανία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Λιμπάτσκα. Εκτιμώ ιδιαίτερα αυτά που είπατε για ελλείψεις ε, στην ε, βιομηχανική και τεχνολογική πρόοδο. Όμως δεν έχει φτάσει άραγε η στιγμή έτσι ώστε να ζητήσουμε τρόπους για να προάγουμε, να δώσουμε κίνητρα. Δηλαδή έχω κατά νου ότι είναι απαραίτητο να εφαρμόσουμε φορολογικά κίνητρα ε, για να διασφαλίσουμε ότι οι βιομηχανίες ε, θα ενδιαφέρονται περισσότερο στην ε, εφαρμοσμένη έρευνα. Επίσης θα πρέπει να πούμε με μεγαλύτερη σαφήνεια ότι οφείλουμε να αναζητήσουμε και καινοτομίες. Και επίσης επειδή θέλουμε να προβούμε σε μεγαλύτερες επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη θα πρέπει να αποφασίσουμε να υπάρχει ένας περιορισμός, μάλλον να καταργηθεί ο περιορισμός του 3%, ελλείμματος 3% στις επενδύσεις που έχουν σχέση με την έρευνα και την ανάπτυξη. Νομίζω ε, ότι, λέει ο κύριος Φέντελη ε, θα έχουμε πάντα μια συζήτηση για αυτά που έχουμε και όχι για αυτά ε, που θα έχουμε αύριο. Το πιο δύσκολο για τους πολιτικούς είναι οι αστάθμητοι παράγοντες. Τι δηλαδή ε, θα πρέπει να προβλέψουν για τα επόμενα έτη έτσι ώστε να ε, προτρέξουν ήδη σήμερα. Διερωτώμε λοιπόν κατά πόσο υπάρχουν ε, κάποια σχόλια για το τι θα γίνει στο μέλλον όχι μόνο για το τι πρέπει να ενισχύσουμε από αυτά που έχουμε, αλλά και για το τι πρέπει να κάνουμε κατά τις επόμενες δεκαετίες ε, για να ανακάμψουμε σε πάρα πολλούς τομείς όπου η Ευρώπη προηγείται. Σήμερα όμως διαπιστώνεται ότι παρουσιάζει ε, στέρηση. Πρέπει λοιπόν καταρχήν να επανέλθουμε εκεί που ήμασταν. Τι είδου μεταρρυθμίσεις χρειαζόμαστε για να δώσουμε τη δυνατότητα στις ε, βιομηχανίες να ανακάμψουν κατά τις επόμενες δεκαετίες. Η κυρία Τρόγια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να επανέλθω σε ένα θέμα το οποίο κατά την άποψή μου είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή το θέμα που έχει σχέση με τη διαθεσιμότητα των πόρων. Είπατε ότι όσον αφορά ε, την πρόσβαση στην πίστη, Ορισμένες ε, χώρες ε, έχουν πρόβλημα, κυρίως η Ισπανία και η Ιταλία λοιπόν αυτά όσον αφορά την τραπεζική πίστη. Εγώ όμω θέλω να μιλήσω για τη διαθεσιμότητα ε, δημόσιων πόρων. Είπατε ότι στην Αμερική προέκυψε ανάκαμψη γιατί υπήρξαν πολλέ κρατικές επενδύσει στην έρευνα εκτό από τι ιδιωτικέ. Κυρίως ε, σε ε, μεγάλους τομείς τη έρευνας και της τεχνολογίας, του περιβάλλοντο και το καθεξής. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε περισσότερο στην Ευρώπη. Δεν έχω διαβάσει όλε τις εκθέσει, αλλά δεν ξέρω ε, μήπως μπορείτε να δώσετε κάποιες συγκεκριμένες ε, προτάσεις. Επ' αυτού ε, μπορούν να ακουστούν πολλά σημαντικά σχόλια. Επειδή λοιπόν φιδωλοί οι πόροι θα πρέπει να μελετήσουμε εκείνες τις δυνατότητες που μπορούν να λειτουργήσουν ως δυνατότητα μόχλευσης για την αύξηση των πόρων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέρες Γκέρεκ, Κέρεκ, κύριος Γκίρεκ. Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για τη βιομηχανία, καταρχήν θα πρέπει να γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα στην βιομηχανία μεγάλης κλίμακας, με μεγάλα δίκτυα, την επιχειρηματική ε, βιομηχανία και Αυτά όλα από τη μια πλευρά και από την άλλη την τοπική βιομηχανία, την ανεξάρτητη, η οποία ακόμα τουλάχιστον δεν εντάσσεται σε διεθνή δίκτυα. Αυτή η βιομηχανία δεν έχει πρόσβαση σε, ε, σε, σημαντικά κονδύλια και βασίζεται περισσότερο στην τοπική παράδοση και στις ε, τοπικές αγορές. Νομίζω λοιπόν ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Σιλβέστ, για την παρουσίαση σας. Είδαμε τα στοιχεία που μας παρουσιάζεται. Στην σελίδα 86 της έκθεσης όμως αναφέρεται ότι το 25%, το 75% συγγνώμη, της απασχόλησης ε, προέρχεται από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτό είναι και το ποσοστό για την προστιθέμενη αξία. Ενώ στην επόμενη σελίδα λέτε ότι η Ισπανία, οι ισπανικές επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίες δεν έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Και μάλιστα υπήρξε διάσωση των τραπεζών στην Ισπανία που αύξησε το δημόσιο χρέος από το 7% στο 100% του ΕΠ. Το αποτέλεσμα ήταν να κοπούν οι πιστώσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οπότε θέλω να ρωτήσω, εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρξει κάποια μεγαλύτερη πειθαρχία ή να δημιουργηθεί μια δημόσια τράπεζα, μια που οι ιδιωτικές τράπεζες δεν στηρίζουν την ανάπτυξη γιατί δεν στηρίζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστούμε κύριο Σέλμερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μιλήσαμε για τις τιμές ενέργειας και μιλήσαμε επίσης και για την επαναγκατάσταση επιχειρήσεων στην Αμερική. Ε, θα συμφωνήσετε άραγε μαζί μου ότι χάσαμε όμως την ουσία. Η ουσία είναι ότι αυτή η επαναγκατάσταση των επιχειρήσεων έχει προχωρήσει ταχύτατα στην Αμερική. Γιατί εκεί υπάρχει το πλεονέκτημα των ιδιαίτερα ανταγωνιστικών ενεργειακών τιμών και η επαναγκατάσταση των επιχειρήσεων στην Ευρώπη προχωράει ανταυτού ε, πολύ αργά διότι έχουμε επιτρέψει τον εαυτό μας ιδιαίτερα υψηλές ενεργειακές τιμές. Με τον τρόπο αυτό υπονομεύσαμε την ανταγωνιστικότητά μας, άρα δηλαδή χρειαζόμαστε νέες πολιτικές για να αντικαταστήσουμε τις αποτυχημένες τις παλιές. Πρόεδρος, αγαπητοί συνάδελφοι, όπως βλέπετε το θέμα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και εγώ προτείνω την ε, ψηφοφορία να την καθυστερήσουμε για 15 λεπτά διότι έχω άλλου, άλλους έξι συναντέλφους στον κατάλογό μου και πρέπει να ακούσουμε και τις απαντήσεις από την εισηγήτρια. Αν ε, λοιπόν συμφωνείτε να αρχίσει η ηλεκτρονική ψηφοφορία με καθυστέρηση 15 λεπτών, γιατί από ό,τι φαίνεται ε, το θέμα που συζητάμε είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε και τον κύριο Τούρμες εκ μέρους των Πρασίνων και τον κύριο Ρούμπεκ, μάλλον ο κύριος Ρούμπι και θέλει ε, να πει κάτι διαδικαστικό. Κοιτάξτε, παρόλα αυτά να γίνει η ψηφοφορία στις 10 ε, και μετά τη ψηφοφορία να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα να ψηφίσουμε τώρα και μετά να συνεχιστεί η συζήτηση. Πρόεδρος δυστυχώς εκτός μικροφώνου. Κοιτάξτε, εφόσον ε, προτείνετε αυτό που προτείνατε, συμφωνώ, αλλά μην ξεχνάτε ότι μερικές φορές ε, οι ομιλητές μας δεν έχουν χρόνο και δεν είναι πάντα εύκολο να γίνεται κάτι τέτοιο. Αν όμως θέλετε να ψηφίσουμε, μπορείτε εσείς να περιμένετε, εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα, μπορεί να περιμένει η συγγήτρια. οι συντονιστές να εξετάσουν αυτό το πρόβλημα, πώς θα το αντιμετωπίζουμε. Εντάξει, σήμερα ας γίνει ψηφοφορία στις 10, γιατί πολλοί συνάδελφοι μπορεί να μην έχουν χρόνο πάνω από 20-25 λεπτά και βεβαίως και είναι απόλυτος απαραίτητο ε, να είσαστε παρόντες κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας της συνεδρίας των συντονιστών. Θα το εξετάσουμε αυτό το πρόβλημα. Εντάξει, ξέρουμε ότι για σήμερα η ομιλήτρια δεν έχει πρόβλημα. Αν θέλει μπορεί να πιει κι άλλο λίγο τσάι για να περάσει η ώρα της. Λοιπόν, ψηφίζουμε. Full agreement.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 ε, Ο κύριος Μπόνι αντικαθιστά τον κύριο Λεβαντόφσκι. Ο αριθμός θα πρέπει να είναι σωστός. Με αυτόν που ψηφίζουν, έτσι. Ωραία. Οπότε αρχίζουμε. Το θέμα είναι Γενικός Προπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015. Όλα τα τμήματα. Αγαπητοί συνάδελφοι, αν έχετε κάποια παρατήρηση στα χαρτιά σας που λέει ότι η ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά πρέπει να έχετε τις κάρτες σας μαζί. Γιατί βλέπετε κάθε τόσο πρέπει να ελέγχουμε ένα αποτέλεσμα, γιατί δεν είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να δούμε διανατάσεις στους χειρών. Και η τελική ψηφοφορία πάντα γίνεται ηλεκτρονικά. Συνεπώς, μην το ξεχνάτε παρακαλώ αυτό στο μέλλον. Οπότε, ψηφίζουμε. Όπως βλέπετε, έχουμε διάφορες τροπολογίες με τέσσερα νούμερα, είναι πολλές. Εγώ θα διαβάζω μόνο τα δύο τελευταία νούμερα. Δεν θα λέω ας πούμε 5906, θα λέω 06 μόνο. Μετά 00 θα λέω ή 01. Γιατί νομίζω είναι αναγνωρίσιμες έτσι οι τροπολογίες χωρίς πρόβλημα και θα είναι πολύ πιο εύκολο να καταλάβουμε τι ψηφίζουμε. Και βέβαια θα λέω υπέρ κατά αποχές. Έτσι είναι απλοί οι κανόνες. Τροπολογία 06 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 00. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 01. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 99. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αποσύρεται εκείνη του κύριου Ρούμπεκ. Και πάμε στην 94, τα Γιάννη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 0-0. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 95 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 0-1 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 60 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 02 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 07 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 92 03. Υπέρ, Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 09 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ρούμπικ και Μπούζικ μαζί τροπολογίες υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. 05. Τροπολογία Μπούζεκ. Α, ε, του Ταγιάννη αποσύρθηκε. Αποσύρθηκε. Συγγνώμη που δεν σας το πω. 05 λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 97 υπέρ κατά, αποχές, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίστε. Εγκρίνεται. Μηδέν. 7 και την 1H. Ε, Τριάντα υπέρ 16 κατά. Εγκρίνεται σαφώς. μηδεν επτά δεκαοχτώ υπέρ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. No H. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 0,9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 08 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ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 και 23 μαζί. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 28 και 24 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 29 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 30 και 25 μαζί υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 31 και 26 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 11 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τώρα πάμε στην 32 και 27 μαζί υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 33 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 12. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ ε, κατά αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 39 και 28 μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 40 και 29 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 41 και 30 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 42, 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 43 και 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 44 και 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 45 και 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 46 και 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 47 και 36 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 48 και 37 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 49 και 38 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 50 και 39 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 98 υπέρ, κατά, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Μπορείτε να ψηφίσετε. 59-98, έτσι. Έχουμε ένα παραπάνω από την Άλντε. Και δύο από το ΕΛΚ παραπάνω. Και ήμασταν έτοιμοι να ψηφίσουμε. Λοιπόν, για να αλλάξει αυτό. Άλντε και ΕΛΚ. Εντάξει είναι τώρα. Πέρα στις ψηφοφορίες. Το αποτέλεσμα το βλέπετε. Εγκρίνεται. 0,6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Να ελέγξουμε θέλετε. Ωραία, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Μπορείτε να ψηφίσετε. Ψηφίσατε όλοι. Τι έγινε, έχουμε παραπάνω από το Και δύο από τους σοσιαλιστές παραπάνω. Θεέ μου, σας αρέσει να ψηφίζετε, δεν το ξέρα, λέει ο πρόεδρος. Έχουμε ένα σοσιαλιστή παραπάνω. εντάξει. Τώρα είναι εντάξει. Α, και έναν από το ΕΛΚ. Εγκρίθηκε. 51. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 και 53 μαζί. Όχι. Μόνο την 14, όχι μαζί λοιπόν. Μόνο η 14. Ψηφίζουμε χωριστά. Είχα μια λαθασμένη πληροφορία εδώ. 14 λοιπόν. Υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 04 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 05 υπέρ, κατά αποχές να ελέγξουμε εδώ. 05. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Μπορείτε να ψηφίσετε. Ψηφίσατε όλοι και παραπάνω όπως θα έπρεπε. Το ΕΛΚ έχει έναν παραπάνω ακόμα. Ψηφίσατε όλοι. Εντάξει είναι τώρα. Εγκρίθηκε. Τσίμα τσίμα το αποτέλεσμα. 57 και 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 58 και 41 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 59 και 42 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 60 ε, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 61 και 43 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. 62 και 44 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. 63 και 45 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται, 64 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 65 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 66 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 67 και 46 μαζί υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται, 68 και 47 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται, 69 και 48 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται, 70 και 49 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. 71 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 72 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 73 και 50 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. 74 και 51 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 76 και 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 77 και 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 78 και 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 81 υπέρ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 παραπάνω από όσους πρέπει να έχουμε από τους σοσιαλιστές. Για την 0-2 ψηφισμό, έτσι τώρα είναι εντάξει. Εγκρίθηκε 0-3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε και για την 0-3. Μπορείτε να ψηφίσετε. ΕΛΚ. Α, όχι, τώρα εντάξει ψήφισατε. Εγκρίθηκε. 90 τώρα. 90 υπέρ. Υπήρξε ένα τεχνικό πρόβλημα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Λοιπόν, ψηφίσαμε ηλεκτρονικά για την 03. Αποτέλεσμα. ...33 ψήφοι υπέρ, 25 ψήφοι κατά και δύο αποχές. Το βλέπουμε εμείς στην οθόνη μας, δεν μπορείτε εσείς να το δείτε στην οθόνη σας, δεν ξέρω γιατί, κάποιο τεχνικό πρόβλημα. τις μικρές οθόνες φαίνεται. Ε? Α, εντάξει, άρα κάνα πρόβλημα. 9-0 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 91 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 92 και 57 μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 93 και 58 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Τελική ψηφοφορία τώρα που θα γίνει ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Τρεις παραπάνω το ΕΛΚ. Μεγαλώνεται. Όλο και περισσότεροι. Α, εντάξει. Ένας παραπάνω ακόμα. Τώρα είναι εντάξει. Αποτέλεσμα. 45 υπέρ, Πέντε κατά και 11 αποχές. Συνεπώς, τελειώσαμε με αυτήν την περίπλοκη κάπως ψηφοφορία και τώρα έχουμε μια πάρα πολύ σύντομη Είναι η δεύτερη ψηφοφορία που έχουμε εδώ και έχει να κάνει με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Επιτρέψτε μου εδώ να σας ενημερώσω για το εξή, γιατί είναι τόσο σημαντική δηλαδή αυτή η ψηφοφορία. Για τη βάση του άρθρου 73, πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής πρέπει να υπερψηφίσουν την τροποποίηση της διαπραγματευτικής ομάδας που θα υιοθετηθεί. Συνεπώς, 33 ψήφοι απαιτούνται. Θα ψηφίσουμε έτσι καλώς ηλεκτρονικά. Χρειαζόμαστε λοιπόν 33 34, 34, πλειοψηφία γιατί έχουμε 67 μέλη στην Επιτροπή μας. Άρα με 34 περνάει. Φυσικά περιμένουμε ακόμα τη θέση του Συμβουλίου, την εντολή. Αλλά εμεί πρέπει να είμαστε έτοιμοι ως Κοινοβούλιο από πριν. Θέλω λοιπόν να σας υπενθυμίσω, που και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην προηγούμενη θητεία του ενέκρινε την θέση του σε πρώτη ανάγνωση και η απόφαση της Επιτροπής μας, της νέας Επιτροπής Ήτρε, της 22ης Ιουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 229 του κανονισμού, επιβεβαίωσε την ε, θέση μας σε πρώτη ανάγνωση της προηγούμενης θητείας. Εσείς το αποφασίσατε αυτό, εσείς το επιβεβαιώσατε αυτό δηλαδή. Συγχρόνως η κυρία Τελκαστήγιο επιβεβαιώθηκε στη θέση της εισηγήτριας για το θέμα αυτό. Ήταν εισηγήτρια και στην προηγούμενη θητεία. Συνεπώς τώρα ψηφίζουμε για την εντολή, τη διαπραγματευτική εντολή τη διαπραγματευτική ομάδα. Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ο πρόεδρος της Επιτροπής, και σκιώδη συγητής, ίσως και κάποιοι άλλοι, βάσει του άρθρου 54. Συνεπώς δεν πρόκειται για καμιά πολύ μεγάλη ομάδα. Και σας υπενθυμίζω, που και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι η Ιταλική Προεδρία θεωρεί προτεραιότητα το θέμα αυτό. Και έτσι ετοιμάζονται και αυτοί ώστε όσο γίνεται πιο γρήγορα να προχωρήσουμε. Εμείς όμως είμαστε πριν από αυτούς και θα είμαστε καλά προετοιμασμένοι για την διαπραγμάτευσή μας. Είμαστε έτοιμοι εφόσον ψηφίσουμε για τη διαπραγμάτευση και για τη σύνθεση της διαπραγματευτικής μας ομάδας, πράγμα που θα κάνουμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Συνεπώς, Αντιλαμβάνομαι ότι όλα είναι σαφή, σωστά. Ας ψηφίσουμε λοιπόν. Μπορείτε να ψηφίσετε ηλεκτρονικά. Πέρα στις 55 υπέρ, 2 κατά. Τέσσερις αποχές. Οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Επόμενη, μάλλον η ομιλήτριά μας εδώ πέρα, μετά από δύο καφέδες, τσάγια, τι ήταν. Τώρα είσαστε σίγουρα σε πολύ καλύτερη κατάσταση, οπότε ελάτε και πάλι για να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Αν κάποιος θέλει να βγει από την αίθουσα, παρακαλώ, όσο γίνεται πιο γρήγορα. Θέλουμε βέβαια να σας κρατήσουμε όλους εδώ στην αίθουσα μαζί μας. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μείνετε στην αίθουσα μαζί μας κι άλλο, αλλά τι να κάνω. Ωραία. Ας ολοκληρώσουμε την συζήτηση που είχαμε αρχίσει πριν την ψηφοφορία. Καθίστε παρακαλώ όλοι στις θέσεις σας πάλι. Ας αρχίσουμε. Ο κύριος Τουρμές θέλει να μιλήσει εκ μέρους των Πρασίνων, σωστά? Γιατί δεν ακούσαμε τη θέση σας πριν. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ένα ερώτημα έχω. Διάβασα τα συμπεράσματά σας εντάχει. Αληθεύει ότι στις χώρες εκείνες, όπως παραδείγματος χάρη η Δανία, που οι τιμές της ανέργειας είναι σχετικά υψηλές, το γεγονός ότι είναι ακριβώς, ε, ιδίως για το ρεύμα, υψηλές οι τιμές, αυτό έχει τη θετική έκβαση ότι οι βιομηχανία όπως δείχνουν και τα στατιστικά στοιχεία είναι πιο αποδοτικοί. Δηλαδή, ο συνδυασμός πραγματικών τιμών με πλήρως ε, εσωτερικευμένο το εξωτερικό κόστος, συν συγκεκριμένα προγράμματα χρηματοδότησης ε, των κυρωτών βιομηχανιών, έχει ως αποτέλεσμα μια πιο ανταγωνιστική βιομηχανία σε σχέση με τις χώρες εκείνες που προσπαθούν να δώσουν στη βιομηχανία τεχνητά φθηνότερο ρεύμα και παραμελούν την ενεργειακή απόδοση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπουτικόφερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να εστιάσω σε μία μόνο πτυχή της έκθεσης και συγκεκριμένα την ανέφεραν και άλλοι συνάδελφοι, την πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Πρέπει να σας πω ότι διαβάζοντας τα πορίσματα σε σχέση με την εμπειρία των ΜΜΕ, αυτό είναι το βασικό τους πρόβλημα και βέβαια και εξέβρεση πελατών. Με βάση τα στοιχεία σας είναι το σημαντικότερο από όλα τα άλλα ζητήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Είμαι λοιπόν λίγο απογοητευμένος, διότι δεν βλέπω στη μελέτη να διατυπώνονται αρκετές προτάσεις για το πώς μπορεί να αλλάξει αυτή η κατάσταση και να σας πω ότι η Επιτροπή μας μόλις τώρα ψήφισε κατά δύο προτάσεων που θα αύξαναν τη χρηματοδότηση για την καινοτομία μεταξύ των μείων. Δυστυχώς. Υπήρξαν ιδέες πάντως, συζητήθηκαν ευρέως, αναφέρεται την ασφάλεια, αλλά δεν αναφέρεται την αξιοποίηση των περιφερειακών κονδυλίων ή τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις ή ομαδικές εξαιρέσεις για μηχανισμούς μερικής ε, απόδοσης ε, κτλ. Πολλές είναι ιδέες που υπάρχουν. Οι αγορές ομολόγουν για περιφερειακές ΜΜΕ. Δεν είμαστε τόσο φιλόδοξοι ε, ως προς την αντιμετώπιση του πολύ σημαντικού αυτού προβλήματος. Ευχαριστώ, λέω πρώτος κύριε Γκροστέτ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Διότι η κυρία Σιλβέστ μας παρουσίασε όλους τους όρους που είναι απαραίτητοι για την ανάκαμψη μέσω της βιομηχανίας όμως. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών μας, έχω το εξής ερώτημα. Ποια είναι τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να ευνοηθεί η βιομηχανική ανταγωνιστικότητα. Έχουμε κάνει λόγο για όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη βιομηχανική ανάπτυξη, όμως δεν έχει γίνει λόγος για την Ευρωπαϊκή Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων. Τι είναι κατεπήγον λοιπόν να αποφασιστεί ώστε να μπορέσουμε να ευνοήσουμε την βιομηχανική ανταγωνιστικότητα. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ηλικιώτης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, τα τελευταία χρόνια γίνεται μεγάλη συζήτηση ότι πρέπει να υπάρξει στροφή στην πραγματική οικονομία για τη δημιουργία θέσεων εργασίας αλλά και για να μπει ε, οι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε ανάπτυξη. Δεν βλέπουμε όμω να υπάρχουν αρκετά μέτρα και ιδιαίτερα θα έλεγα για τον Νότο που συμφωνώ με προηγούμενου συνάδελφου βρίσκεται σε μια διαδικασία αναποβιομηχανοποίηση να υπάρχουν αρκετά μέτρα στήριξη σε αντίστοιχο που υπάρχει ε, για στήριξη του τραπεζικού τομέα ε, και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Άρα ε, χρειάζεται να, έχουμε, να δούμε, και εδώ θέλω την απάντηση σας, μια πιο συγκεκριμένη πολιτική σε ό,τι αφορά τη στήριξη της βιομηχανίας και των μικρομεσών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στην Νότια Ευρώπη. Το δεύτερο, το 2012 ξεκίνησε μια συζήτηση στο πλαίσιο και της Επιτροπής και του Συμβουλίου ε, για το θέμα των κρατικών ενισχύσεων. Είναι αλήθεια ότι για να μπορέσουν η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να ανταγωνιστεί με επιτυχία ε, άλλες χώρες πρέπει να ξαναδεί ε, σε μεγάλο βάθος το ζήτημα των κρατικών ενισχύσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των, ε, στην Ευρώπη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Thank you Ευχαριστώ κύριος Λάμστορφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το πιο κατεπήγον νομίζω είναι να σταματήσω πάλι στην Ουκρανία για να λυθούν τα προβλήματα για τα οποία συζητούμε σήμερα. Υπάρχει ο κίνδυνος ε, να έχουμε μια τεχνική αστοχία της Κεντρικής Τράπεζας στην ε, περιοχή αυτή μια ε, στάση πληρωμών. Για να το αποφύγουμε αυτό πρέπει να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, να σταματήσει ο πόλεμος. Το δεύτερο, η απειλή της ενεργικής κρίσης στην Ουκρανία είναι ένα μεγάλο θέμα, διότι σε 40 ημέρες θα έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα ε, έλλειψης, παράδοση ενέργειας ηλεκτροδότηση δηλαδή για τους πολίτες και ε, παροχή ηλεκτροδότηση για τις βιομηχανίες. Θα έχουμε πρόβλημα. Είναι κρίσιμη κατάσταση. Δεν υπάρχουν λύσεις. Αναφέρθηκε η αποψήλωση δασών, η χρησιμοποίηση υπερτομάτων ζώων και άλλα ε, θέματα. Όχι, δεν θα λύσουν το πρόβλημα πρέπει με τη διεθνή συμβολή να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. Γιατί αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα πάρα πολύ μεγάλα βάρη και για πολλά χρόνια για την οικονομία της Ευρώπης. Ähm, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν πάρα πολλέ καλέ παρατηρήσει σε αυτή τη μελέτη, αλλά θα ήθελα να φερθώ σε κάτι που είπε ο κ. Πιουτικόφερ. Δηλαδή, τελικά αν οι πράσινοι αποδίδουν τόσο μεγάλη σημασία στα διαρθρωτικά ταμεία και υποτίθεται σε πολλά που δεν περιλαμβάνει η μελέτη, τότε εγώ θέλω να σας πω το εξής. Μία ενίσχυση εγκατάστασης ε, που καταβάλλεται στη Νότια Ευρώπη, αυτή καταβάλλεται μόνο εφάπαξ και ε, μετά την έντρα που έχει η εταιρεία την έχει για τουλάχιστον τα επόμενα 10-20 χρόνια. Άρα δηλαδή είναι πολύ πιο σημαντικό να υπάρχουν ενεργειακές υποδομές, σωστή εκπαίδευση, σωστές αγορές, ε, δυνατότητες μεταφοράς και για όλα αυτά τα θέματα υπάρχουν πάρα πολύ καλές προτάσεις στη μελέτη σχετικά με τις υποδομές. Βεβαίως και για μένα κάτι λείπει και αυτό είναι η άδικη μεταχείριση των επενδυτών. Αν στη Νότια Ευρώπη έχω την ίδια ιδέα όπως στη Γερμανία ή στην Πολωνία, τότε ξέρετε στη Νότια Ευρώπη δυστυχώς το κόστος των δανείων ε, είναι διπλάσιο για την ίδια επιχειρηματική ιδέα. Και αυτό κατ' ουσίαν είναι το μεγάλο μας πρόβλημα, ότι την πολιτική χαμηλών επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν μπορούμε να την διοχετεύσουμε στην πραγματική αγορά. Άρα δηλαδή για την Νότια Ευρώπη, για μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να περιορίσουμε το ε, κόστος το πιστοτικό. Δεν μιλάω για νέα προγράμματα, αλλά μιλάω για δάνεια τα οποία χορηγούνται από τις τράπεζες. Και νομίζω ότι αυτό πραγματικά είναι το πρώτο καθήκον και μέλημά μας και βλέπω ότι δεν υπάρχει. Ο κύριος Ταγιάννη. Πρόεδρε, εγώ πιστεύω ότι αυτή η μελέτη είναι σημαντική, διότι επιτέλους ε, μετά από όλο αυτό το καιρό αρχίσαμε να μιλάμε για τη βιομηχανική πολιτική. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι για να υπάρξει μια νέα βιομηχανική πολιτική θα πρέπει να κάνουμε αυτό που κάναμε ήδη κατά την προηγούμενη θητεία του Κοινοβουλίου και το έκανε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή εγκρίναμε μια στρατηγική ε, βιομηχανικής ε, πολιτικής, ε, υπήρξαν επενδύσεις περίπου 10 δις στην πραγματική οικονομία για να υπάρξει μια ουσιαστική βιομηχανική πολιτική έτσι λοιπόν ορισμένες απαντήσεις στις ερωτήσεις που έκαναν οι συνάδελφοι περιλαμβάνονται ήδη στο έγγραφο της Κομισιόν ε, για τη στρατηγική της. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση και κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας να εκμεταλλευτούμε τη δουλειά μιας επιτροπής ε, της οποίας ε, προείστατο ένας ε, πρόεδρος, ο οποίος παλιά ήταν και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Άρα δηλαδή η φωνή αυτής της Επιτροπής είναι κάπως πιο ισχυρή και δεν πρέπει απαραίτητα να επιλέξουμε η βιομηχανική πολιτική να ασκείται μόνο από το Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο και αυτό πρέπει να το δείξουμε και στις ακροάσεις που θα κάνουμε στους επιτρόπους ε, το θέμα ας πούμε του Επιτρόπου για την Οικονομία. Σε αυτόν επιμείνουμε στην ε, πραγματική βιομηχανία. Εγώ λοιπόν προτείνω παράλληλα με το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ να υπάρχει και ένα Συμβούλιο που να λέγεται της πραγματικής οικονομίας γιατί αυτό το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας ε, τελικά κινδυνεύει να καταλήξει μόνο σε ένα Συμβούλιο των Πρέσβεων. Αυτό που ενδιαφέρει είναι τα μακρο και μικροοικονομικά να τα φέρουμε σε κάποια ισορροπία και έτσι λοιπόν το Κοινοβούλιο μπορεί να οδηγήσει στην ύπαρξη ενός ε, Συμβουλίου Πραγματικής Οικονομίας παράλληλα με το Συμβούλιο Σας ευχαριστώ πολύ. Έχετε μεγάλη εμπειρία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σίγουρα αυτό θα βοηθήσει τα μάλα στη διατύπωση των ιδιών αυτών που θα μπορούσαν έπειτα να εφαρμοστούν στο Κοινοβούλιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ολοκληρώνουμε λοιπόν τον κατάρα τον για το τελευταίο τη δεν θέλει το λόγο και σα δίνουμε το λόγο για να δώσετε τι απαντήσει σα. Θα ήθελα να σα πω αγαπητοί συνάδελφοι ότι την επόμενη φορά θα έχουμε τον ε, Επίτροπο Φερότσι για το θέμα αυτό ακριβώ. Ανταγωνιστικότητα τη Ευρωπαϊκή οικονομίας και επαν Ο κ. Φερότσι λοιπόν Επίτροπος θα, συζητηθεί, θα συζητήσει μαζί μας αυτό το θέμα. Άρα σε καμία περίπτωση δεν λύγει σήμερα αυτή η συζήτηση. Κύριε Κρίφαν, θέλετε να πει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλή είναι η ανάλυση, αλλά τι κάνουμε. Μιλήσαμε ε, για την πρόσβαση στην ανάπτυξη σε ε, διάφορους τομείς η αυτοαπασχόληση όμως που δεν αναφέρεται, ιδίω στον Ηνωμένο Βασίλειο, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ίσω και για να καλύψει χαμηλά αμοιβόμενε θέσει εργασία. Πώς θα δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον για καλή, για ποιοτική αυτοαπασχόληση σε τομεί ψηλή ανά, και τι κάνουμε ώστε η επιταχυμένη μαθητεία να προωθηθεί ακόμη περισσότερο. Ωραία. Θα δώσω και στην κυρία Μπερέ όμω το λόγο. Είναι η τελευταία και δεν υπάρχει καμία άλλη, κανένα άλλο που θα ακολουθήσει. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση γύρω από την ε, μελέτη αυτή που κάνατε είναι πολύ σημαντική και πλούσια στην αρχή αυτής της κοινοβουλευτικής θητείας. Εμάς ε, βέβαια μας απασχολεί πολύ και η συγκρότηση της επόμενης Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα παρατηρήσατε ότι όταν ήταν αρμόδιος για τα βιομηχανικά ζητήματα ο κ. Σταγιάννη στην προηγούμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, πώς ε, αντιμετωπίζονταν αυτά τα ζητήματα, πώς, ποιες είναι οι πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τώρα αυτά τα θέματα, τι συντονισμός μεταξύ των χαρτοφυλακίων θα υπάρξει για να υπάρχει μια ευφυής αντιμετώπιση των στρατηγικών αυτών. Ευχαριστώ. Έχετε το λόγο. Οριστικά πια. Δικό σας ο λόγος. Μάλιστα. Να κάνω μια ομαδοποίηση των ερωτήσεων. Μου υπενθυμίσατε καταρχάς ότι δεν απάντησα στο ερώτημα για το τι μπορεί να γίνει με την επανεγκομηχάνηση στην Νότια Ευρώπη. Είναι ένα θέμα. Έχουμε ήδη πολλά εργαλεία σε ισχύ, τα διαθετικά ταμεία για τη χρηματοδότηση των υποδομών, αλλά και χρηματοδότηση προγραμμάτων ε, απευθείας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αξιοποίηση, μέγιστοποίηση των διαθέσιμων πόρων για να βοηθηθεί η βιομηχανία στην Νότια Ευρώπη. Και ιδίως στις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση. Τώρα, το αν πρέπει να τεθεί θέμα κρατικών ενισχύσεων είναι πολιτικό το ζήτημα. Αυτό δεν έχω απάντηση. Τα διαθωτικά ταμεία όμως είναι ένα εργαλείο που υπάρχει και αναμένει την πλήρη του. Υπήρξαν ερωτήσεις επίσης για την καλύτερη διήθμιση, δικτικά προβλήματα, τι μπορούμε να κάνουμε. Η κυρία Καστίγιο, δεν είναι εδώ βέβαια πια, αλλά Ναι, καλύτερη ρύθμιση, νομίζω είναι παρόν αναφέρεται και στην έκθεση, και έχουν γίνει και πολλά ήδη. Σίγουρα πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες, να έχουμε μελέτες αντικτύπου των νέων νομοθετημάτων, ώστε να είναι ελάχιστα ε, τα βάρη προς τις επιχειρήσεις. Πολλά διοικητικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στα κράτη-μέλη οφείλονται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και οξύνεται από την κακή συχνά εφαρμογή από τα κράτη-μέλη. Αν δηλαδή υπήρχε πλήρης εφαρμογή και δεν γινόταν κάτι επαφενειακό, τότε δεν θα ήταν τόσο πολλά τα προβλήματα σε ορισμένα κρατημέλη. Επίσης, υπήρξαν κάποιες ερωτήσεις για τη χρηματοδότηση της καινοτομίας και της έρευνας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω από κοινού στα περισσότερα από αυτά τα ερωτήματα. Φορολογικά κίνητρα για φορολογική ε, πίστη, για την καινοτομία, για την έρευνα και την ανάπτυξη. Υπάρχουν ε, τέτοια κίνητρα. Τώρα σε ποιο βαθμό είναι παρόμοια ή διαφέρουν ε, από κράτος μέλος σε κράτος μέλος, αυτό δεν το γνωρίζω. Κάποια έχουν 100% φοροπαλλαγή για έρευνα και καινοτομία, αλλά λιγότερο. Σίγουρα κάτι μπορούμε να κάνουμε. διδικοσίες διαγωνισμού, προμήθειες, ήδη με το πλαίσιο που έχουμε μπορούν να ληφθούν υπόψη απαιτήσει για την ενίσχυση της καινοτομίας. Στο πλαίσιο λοιπόν των κανόνων για τους δημόσιους διαγωνισμούς μπορεί ε, να υπάρχει αυτή η, η απέτηση, η απαιτησότητα, τεχνολογική καινοτομία. Η χρηματοδοτούν την έρευνα για δημόσιου σκοπού, στρατιωτικό τομέα για παράδειγμα. Είναι πολύ γνωστό αυτό, τα καταφέρνουν πολύ καλά οι Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, έχουν διάφορα προγράμματα κρατική χρηματοδότηση. Και πάλι όμω ε, στο πρόγραμμα για το 2020 έχουμε τέτοια εστίαση και εμείς ή με τις συμπράξεις δημόσιου τομέα ή με την ανάπτυξη συγκεκριμένων νέων τεχνολογιών που είναι προς το δημόσιο συμφέρον. Μάλλον μόνο ένα λεπτό μου έχει απομείνει. Δεν νομίζω ότι μπορώ να απαντήσω όλα τα ερωτήματα. Για την ενέργεια, το ενεργειακό κόστος φυσικά και είναι πρόβλημα. Το θέμα είναι να βρεθεί ισορροπία. Και πρέπει να υπάρξει εξισορρόπηση ε, μεταξύ των διαφόρων πολιτικών. Στη χώρα μου τη Δανία για παράδειγμα. Το υψηλό ενεργειακό κόστο ήταν κίνητρο για τι επιχειρήσει να γίνουν πιο ενεργειακά αποδοτικέ ή αποδοτικές, περισσότερο αποδοτικέ ω προ το κόστο, χρήση πράσινων τεχνολογιών κτλ. Είναι ένα κόστο, ένα μάλλον κίνητρο να γίνουν ενεργειακά πιο αποδοτικέ οι επιχειρήσει, αυτό το υψηλό ενεργειακό κόστο. Αλλά όχι να υπάρχει αυτή η δικαιολογία για να διατηρείται η για ενεργειακού κόστο. Τέλο πάντων, το θέμα είναι πολιτικό. Εγώ δεν μπορώ να διατυπώσω κάποια σύσταση. Θα σα δώσω λίγο παραπάνω χρόνο γιατί δεν θα είναι ευχαριστημένοι συνάδελφοι αν δεν απαντηθούν τα ερωτήματά του, λέει ο Πρόεδρο. Μάλιστα, για να δούμε. I don't think I have an opinion on that. On that. Για <laughs> την επόμενη επιτροπή δεν μπορώ. Δεν μπορώ να εκφέρω άποψη. Υπήρχαν διάφορα ερωτήματα για τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν. Νομίζω δείχνει σαφώς και η μελέτη ότι το θέμα είναι άκρος πολύπλοκο. Πολλά είναι αυτά που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Το ενεργειακό κόστος είναι ένα πρόβλημα αλλά για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σημασία έχει να περάσετε την βελτίωση της λειτουργίας της ε, εσωτερικής αγοράς, πρόσβαση στη χρηματοδότηση, ορίζον 2020, το πρόγραμμα αυτό αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα που έχουν να κάνουν με την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, αλλά μεγάλο βάρος έχουν και ιδιωτικέ αγορές. Θέλουμε να μπούμε στα γρανάζια ε, τη λειτουργία τη εσωτερική αγορά. Αυτό είναι το ερώτημα και αφήνω στους πολιτικού να το απαντήσουν. Πρέπει όμω να έχουμε μια εξισορρόπηση μεταξύ δημόσια στήριξη ε, και ιδιωτικών αγορών. Κάποιο με παίρνει τηλέφωνο. Υπάρχει κάτι άλλο. Κάποια από τα ερωτήματα και τις παρατηρήσεις Παραδείγματο χάρη, πώ θα οργανωθούν τα, ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ε, πώ θα επηρεάσουμε τα κράτη-μέλη, πώ θα προωθήσουμε την επανεβιομηχάνηση, την ενεργειακή απόδοση, τι σημαίνει ενεργειακό κόστο, ανταγωνιστικότητα τη βιομηχανία μα. Φυσικά και θα πρέπει να τα συζητήσουμε αυτά τα προβλήματα και αυτό θα το πράξουμε στην προσεχή μας ε, ε, συνάντηση με τον Επίτροπο Νέλη Φερότσι. Να πω ότι η κυρία Γιάννη Σίλβεστ εκπροσωπεί το Δανέζικο Τεχνολογικό Ινστιτούτο. Μας παρουσίασε μια εξαιρετική έκθεση. Θέλω να σας ε, ευχαριστήσω θερμά κυρία μου. Παρακαλώ χειροκροτήστε συνάδελφοι. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτή. Κυρία μου, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν εδώ μαζί μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε στο επόμενο σημείο. Σημαντικό. Η ανανέωση της εντολής του επιτελεστικού διευθυντή του ΕΝΙΣΑ, δηλαδή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών. Δύσκολα μπορώ να θυμηθώ όλη την ονομασία, αλλά τέλος πάντων ο ενής είναι πολύ σημαντικός. Ξέρουμε πόσο σημαντική είναι η ασφάλεια των πληροφοριών. Πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Ο κύριος Ούντο Χέλμπρεχτ για την ανανέωση της εντολής που θα ε, συζητήσουμε της θητείας του ως εκτελεστικού διευθυντή. Καλώς ορίσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να σας πω ότι για να ανανεωθεί εντολή ε, και η θητεία του εκτελεστικού διευθυντή. Ο υποψήφιο καλείται να προβεί σε μια δήλωση ενώπιον τη Επιτροπής Ήτρε και να δεχθεί τι ερωτήσει των μελών της Επιτροπή Ήτρε. Αυτό θα γίνει λοιπόν στην συνάντησή μας με τον εκτελεστικό διευθυντή είναι σημαντική αυτή η συνάντηση και για αυτούς τους τυπικούς λόγους, ε, αλλά και γιατί θέλουμε να γνωρίσουμε το περιεχόμενο των δράσεών σας. Για μια ακόμη φορά λοιπόν σας καλωσορίζουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας δίνω αμέσω το λόγο. Ελπίζω να μην ξεπεράσετε τα 10 λεπτά γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ευχαριστώ. Κύριε Μπούζεκ, και μέλη της Επιτροπής ΙΤΡΑ. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω ενώπιόν σας και να σας εξηγήσω τι κάνει η ΕΝΙΣΑ για την Ευρώπη. Ονομάζομαι Ούντο Χέλμπερ και τον Οκτώβριο του 2009 ορίστηκα εκτελεστικό διευθυντή. Μέσα στα επόμενα λεπτά θα σα εξηγήσω γιατί είναι σημαντικό ο οργανισμό ΕΝΙΖΑ και τι μένει να κάνουμε. Πρόκειται για έναν ευρωπαϊκό οργανισμό που είναι στο κέντρο των αρμοδιοτήτων όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια στην Ευρώπη. Έχουμε 70 άτομα προσωπικό και 10 εκατομμύρια ευρώ προπολογισμό. Έδρα μας είναι η Ελλάδα. Έχουμε ένα λειτουργικό τμήμα, επιχειρησιακό τμήμα μάλλον στην ε, Αθήνα και διοικητικό προσωπικό στο Ηράκλειο. Από το 2009, το το 2009, η οικονομική διαχείριση έχει βελτιωθεί πάρα πολύ και η ΕΝΗΣΑ είναι σήμερα ένας από τους καλύτερα ε, λειτουργούντες ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Εμείς δουλεύουμε για ένα ανοιχτό και ασφαλή κυβερνοχώρο στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, προσπαθεί να ενισχύσει την κυβερνοασφάλεια και να αποφύγει ε, προβλήματα όσον αφορά την ασφάλεια του χώρου αυτού και συμβάντα. Επίσης, συνεισφέρουμε και στην ανάπτυξη της σχετικής πολιτικής για την ασφάλεια δικτύων στην Ευρώπη. Η μεγαλύτερη δύναμή μας είναι οι δεσμοί που έχουμε με τους διάφορους ε, εμπλεκόμενους. Πρώτα απ' όλα και με τον δημόσιο τομέα αλλά και με τον ιδιωτικό τομέα συνεργαζόμαστε και προτείνουμε λύσεις και δίνουμε συμβουλές βασιζόμενες στη δικιά μας εμπειρία. Εμείς προσπαθούμε ε, να δείξουμε ότι η προσέγγιση μας είναι γενός πολλαπλιαστική όσον αφορά το αποτέλεσμα των δυνατοτήτων που προσφέρονται στις χώρες μέλες. Και πιστεύουμε ότι όλοι έχουν αποφελθούν από μια τέτοια προσέγγιση. Αν κοιτάξουμε το 2010, τότε δεν υπήρχε ε, διαχείριση κρίσεων στην Ευρώπη. Σήμερα όμως το 2014 έχουμε συγκεκριμένες επιχειρησιακές διαδικασίες που δοκιμάζονται μέσω ε, δοκιμών ιδιαίτερα περίπλοκων που γίνονται σε όλες τις χώρες μέλη. Γιατί η δουλειά μας είναι σημαντική τώρα. Η τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών είναι κάτι πολύ βασικό για κάθε σύγχρονη κοινωνία. Ένα ανοιχτό λοιπόν και ασφαλή κυβερνοχώρο είναι κάτι πολύ βασικό για να διατηρηθούν οι αξίε μα, όπω είναι αναφέρονται στο χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων και μεταξύ άλλων είναι και η εσωτερική αγορά. Ε, θα έλεγα ότι τα business model είναι κάτι το οποίο προσφέρει πολλές ευκαιρίες για εγκλήματα στο κυβερνοχώρο. Έτσι λοιπόν η ασφάλεια του κυβερνοχώρου είναι πολύ βασική για να μπορέσουν τα δίκτυά μας υποδομών και πληροφοριών να λειτουργήσουν καλά. Είτε πρόκειται για τις τράπεζες, είτε πρόκειται για την ενέργεια, το νερό, για την, ε, τις παραγωγικές βιομηχανίες και οποιοδήποτε άλλο δίκτυο. Το λεγόμενο ίντερνετ των πραγμάτων είναι επίσης κάτι πολύ σημαντικό που μας απασχολεί τον τελευταίο καιρό θα μπορούμε έτσι από μακριά να μπορούμε να ανάβουμε το φως, τη θέρμανση, οτιδήποτε άλλο στα σπίτια μας. Το e-banking, η ηλεκτρονική εκπαίδευση, η ηλεκτρονική υγεία, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία βασίζονται σε έναν ανοιχτό και ελεύθερο κυβερνοχώρο. Είναι τεχνολογίες αυτές που έχουμε χτίσει σήμερα και οι οποίες θα μας επιτρέψουν να έχουμε στη διάθεσή μας έξυπνες πόλεις μέσα στις οποίες να ζούμε έξυπνα. Θα σα παρουσιάσω μια εισαγωγή του τι κάνουμε σήμερα. Στηρίζουμε την ανάπτυξη πολιτική όσον αφορά τις απειλέ στον κυβερνοχώρο. Επίση, δημιουργία ικανοτήτων σε όλε τι χώρε μέλη. Για παράδειγμα, ε, έχουμε φτιάξει ομάδε, οι οποίε δουλεύουν και πάνω στο ε, cloud computing και όσον αφορά την συνεργασία γίνονται δοκιμές για την προστασία δεδομένων, τον ιδιωτικό βίο, εντοπίζουμε παραβιάσεις που γίνονται και στηρίζουμε τις χώρες μέλη και το Το μόνο σταθερό στον τομέα αυτό είναι ότι τα πράγματα αλλάζουν. Αυτή είναι η μόνη σταθερή αξία θα έλεγα. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς δουλεύουμε πάρα πολύ σε δύο τομείς κυρίως, στο cloud computing αλλά και στα ενεργειακά δίκτυα. Το λογιστικό νέφος λοιπόν, το cloud computing, είναι κάτι που αλλάζει πάρα πολύ τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε οι επιχειρήσεις, τα δίκτυα. Ήδη από το 2009 είχαμε δημοσιεύσει την έκθεσή μας σχετικά με το λογισμικό νέφος. Όντως πρέπει να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα. Νέες υπηρεσίες, νέα business models. Το θέμα λοιπόν της ασφάλειας παίρνει όλο και μεγαλύτερη σημασία κυρίως για τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις οι πάροχοι του λογισμικού νέφους λειτουργούν ε, εκτός ε, του ελέγχου μας και έτσι τέτοια κέντρα μπορούν να βρεθούν οπουδήποτε στον κόσμο, πράγμα το οποίο οδηγεί σε πολλές προκλήσεις και σε πολλά ερωτηματικά. Και φυσικά μπορούν να αποτελέσουν και στόχο για επιθέσεις. Νέες λοιπόν ε, επιθέσεις υπάρχουν που απαιτούν νέες συμφωνίες, νέες πιστοποίησεις και προσπαθούμε λοιπόν έτσι να βελτιώσουμε σημαντικά την ασφάλεια. Ο δεύτερος τομέας στον οποίο θέλω να αναφερθώ είναι το θέμα των ευθειών δικτύων ενέργειας και υποδομών. Οι πολίτες ήδη με τα φωτοβολταϊκά οι ίδιοι είναι σε θέση να δημιουργήσουν ενέργεια. Υπάρχουν επίσης νέα κέντρα σιγά σιγά που δημιουργούνται σε κάθε σπίτι και μετά από μερικά χρόνια όλα τα σπίτια διαθέτουν ένα τέτοιο υπολογιστάκο και με λογισμικό θα τα Αν ε, από μακριά μπορεί κάποιος εγκληματίας να σβήσει τους υπολογιστές αυτούς, ξαφνικά δεν θα έχουμε ηλεκτρισμό ή θα μπορούν να κλέψουν ε, ιδιωτικά δεδομένα προσωπικά δεδομένα. Από τεχνική λοιπόν και στρατηγικής άποψη πολλά πράγματα μπορεί να κάνει ακόμα η ενής οργανισμός ενίσα στον τομέα αυτό των δικτύων και της ασφάλειάς τους. Για παράδειγμα, υπάρχουν νέε προκλήσεις όπως είναι το Industry 4, η βιομηχανία 4. Έπειτα, τα μαζικά δεδομένα δίνουν νέε δυνατότητε και ευκαιρίε και αλλαγέ στη συμπεριφορά μα. Τα μαζικά δεδομένα βέβαια θέτουν και προκλήσεις όσον αφορά την ασφάλεια. Έπειτα η φορητή υπολογιστή και αυτή είναι μια τεράστια πρόκληση όσον αφορά την ασφάλεια των δεδομένων μας. Ε, το θέμα της προστασίας της ταυτότητας των χρηστών. Αν ε, κοιτάξουμε τι αναφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το στόχο του 2020, τότε πράγματι ο ΕΝΗΣ έχει να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Επίσης, η εσωτερική αγορά για ε, προϊόντα ασφάλειας και υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαπέτει από ισορροπία. Διότι η αγορά στη... κυριαρχείται από αμερικανικές εταιρείες οι οποίες τονώνουν την προσφορά πολύ περισσότερο από ό,τι να αυξάνουν τη ζήτηση. Ο ΕΝΙΣΑ λοιπόν μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο και στα θέματα της τυποποίησης. Ήδη έχω υπογράψει ένα μνημόνιο κατανόησης με το ΣΕΡΤ ο ΕΝΙΣΑ λοιπόν συνεργάζεται πολύ με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε, όπως σας είπα, υπογράψει το Μνημόνιο Κατανόησης και προχωράμε και σε θέματα νομοθεσίας, κάνουμε προτάσεις για ρυθμίσεις όσον αφορά την ηλεκτρονική ταυτοποίηση. Ας δούμε τώρα ποια είναι τα οράματά μας και η στατική μας στόχη για τα επόμενα χρόνια. Το όραμά μας είναι να χρησιμοποιήσουμε τις μοναδικές ε, ε, τα μοναδικά προσόντα που διαθέτουμε για να βοηθήσουμε στην ασφάλεια δικτύων και πληροφορών. Στην ομοθετική διαδικασία, στην διασφάλιση της ε, κοινωνίας των πληροφοριών και να συνεισφέρουμε επίσης στην ανάπτυξη της ε, ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς. Αυτά θα στηριχθούν με τους εξής στρατηγικούς στόχους. Πρώτον, ε, με την ανάπτυξη και την διατήρηση υψηλού επίπεδου εμπεριγνωμόνων από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα λαμβάνουν υπόψη τις εξελίξεις στην ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών. Δεύτερον, να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην οικοδόμηση ικανοτήτων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτον, να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών που είναι αναγκαίε για να αντιμετωπιστούν οι απαιτήσει από την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών. Και τέταρτον, να ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ χώρων αλλά και μεταξύ ε, περιφερειών. Και θα καταλήξω με εξή. Πιστεύω ότι ο Ενίζα έχει την πραγματογνωμοσύνη που χρειάζεται στον κυβερνοχώρο για να βοηθήσει την Ευρώπη και να αντιμετωπίσει τι προκλήσει αυτέ. Ο Ενίζα τα επόμενα πέντε χρόνια θα δουλέψει με του διάφορου φορεί για να ενισχύσει και τα αποτελέσματα και να φροντίζει να γίνουν οι καλύτερε δυνατών ε, αποφάσει στον τομέα των επενδύσεων. Είπαν νωρίτερα ότι η εντολή μας εκπνέει το 2020 και σύμφωνα με τον κανονισμό μέχρι τις 20 Ιουνίου 2018 η Επιτροπή θα ζητάει αξιολογήσεις από τον οργανισμό μας. Μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια λοιπόν ο ΕΝΙΖΑ αντιμετωπίζει ένα νέο τοπίο που δεν γνωρίζουμε ακόμα, όπου τα δίκτυα πρέπει να είναι περισσότερο ασφαλή από ποτέ και μέχρι το 2018 να βοηθάει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις ανακοινώσεις της και με την νομοθετική διαδικασία να βοηθάει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Πιστεύω ότι ο οργανισμός μας έχει την πλήρη σας υποστήριξη και ελπίζω ότι θα συνεχιστεί αυτό για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος τα επόμενα πέντε χρόνια. Θέλω και να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας, την Ήτρα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γενικότερα για την στήριξή σας και προσβλέπουμε σε καλή συνεργασία προκειμένου να σας εξυπηρετήσουμε και τα επόμενα πέντε χρόνια. Θα κάνω ό,τι μπορώ στο οργανισμό ΕΝΙΣΑ να ανταποκριθεί στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ε, Mr. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Διευθυντά, τηρήσατε το χρόνο σας. Δίλεπτες θα είναι οι παρεμβάσεις ε, των εκπροσώπων των πολιτικών επιτροπών. Από το έλκο κύριος Μπόνι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Διευθυντά, καταλαβαίνουμε όλοι τον αυξανόμενο ρόλο της ασφάλειας και τις προκλήσεις με τις ε, ψηφιακές εξελίξεις που είναι καταιγιστικές. Από την άλλη πλευρά, νέες μορφές επιθέσεων παρατηρούνται, hacking, επιθέσεις, πολλές απειλές στον τομέα του cloud computing που αναφέρατε, στα ενεργειακά δίκτυα, στο ταπεζικό σύστημα, προστασία δεδομένων εν γέν, προστασία δηλαδή ιδιωτικότητας και στο μέλλον το συστήματα ηλεκτρονικής υγείας. Ο ΕΝΙΖΑ είναι πολύ σημαντικός οργανισμός και είναι το μόνο εργαλείο για την αντιμετώπιση των απειλών αυτών. Επομένως, θα πρέπει να υποστηρίξουμε τη δημιουργία ενός καλύτερου πλαισίου για τον ΕΝΙΖΑ και την ανάπτυξή του και καλή νομοθεσία. Έχω ορισμένε ερωτήσει. Πρώτον, Υλοποίηση της οδηγίας για την ασφάλεια των δικτύων και πληροφοριών. Εφαρμόζεται αυτή η οδηγία. Ποια είναι τα εμπόδια που πιθανώς προέρχονται από ορισμένα κράτη-μέλη. Υπάρχει απειλή εφαρμογή τη οδηγία αυτή. Δεύτερον, τι είδου υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρείται ότι θα ήταν χρήσιμη ώστε η οδηγία αυτή να γίνει ένα πραγματικό εργαλείο για να ξεκινήσει μια ανοιχτή ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών μεταξύ εμπλεκομένων μερών και ενδιαφερομένων από τα κράτη-μέλη. Τρίτον, πώς εκτιμάται το ρόλο της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, της εν δηλαδή για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών και την πρόταση για την ε, τροποποίηση του κανονισμού περί προστασίας δεδομένων και ηλεκτρονική αναγνώριση ηλεκτρονικές συναλλαγές στην ιστορική αγορά. Αν τα νομοθετήματα αυτά θεωρείται ότι θα βελτιώσουν την κατάσταση και πώς θα αλλάξει ο ρόλος ε- του ΕΝΙΖΑ με αυτά τα νέα νομοθετήματα. Τέταρτον, τι είδου θεσμική υποστήριξη χρειάζεστε τα επόμενα χρόνια, όπου θα πρέπει να εστιάσετε στην έγκαιρη προεδοποίηση και εντοπισμό νέων προβλημάτων στον τομέα της ασφάλισης. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Έχω ένα τελευταίο ερώτημα. Μπορείτε να πείτε κάτι περισσότερο για αυτό το πολύ ωραίο, όπως ακούγεται τουλάχιστον, ασφάλεια από το σχεδιασμό. Security by design. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ, αλλά παρακαλώ, επειδή δεν έχουμε χρόνο, οι υπόλοιποι να μην μακρηγορήσουν τόσο πολύ. Η κυρία Ντάλι από τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τον εκτελεστικό διευθυντή για την παρουσίασή του και για την έκθεση που τη διάβασα έτσι κάπως πιο αναλυτικά. Εμείς πιστεύουμε ειλικρινά ότι μέσα σε πολύ λίγο χρόνο έχει κάνει σημαντική συμβολή στην ασφάλεια δικτύων πληροφοριών η, ο Ενίζα. Όμως είναι σημαντικό ότι αν συνεχιστεί με την ίδια μορφή, ο οργανισμός αυτός να ισχύει, να υφίσταται, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τον συνεχώ μεταβαλλόμενο κυβερνό χώρο. Μιλήσατε για πόσες αλλαγές βιώνουμε στον κυβερνό χώρο. Επομένως, καλό θα ήταν να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν οι νέε προκλήσει και αυτέ οι αλλαγέ. Και από αυτήν την έννοια, Πρώτα απ' όλα και κυρίως θέλω να σας ρωτήσω πώς προβλέπετε να συνεισφέρει ο οργανισμός στην ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς. Έχετε εντοπίσει τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο οργανισμός. Έχετε ήδη ένα σχέδιο, ένα πλάνο για να τις αντιμετωπίσετε αυτές τις αλλαγές σκέφτεστε να ξεκινήσετε μια στρατηγική για την αποτελεσματική προστασία των ε, παιδιών που μπαίνουν στο διαδίκτυο και η αγορά για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ασφαλής στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ισορροπημένη γιατί δεσπόζουν ε, οι αμερικανικές ε, εταιρείε και λειτουργίες στην αγορά. Πώς μπορεί ο οργανισμός λοιπόν να βοηθήσει να υπάρξει μια νέα ισορροπία. Πρώτα σε ευχαριστώ. Τηρήσατε και το χρόνο σας. Κυρία Έρνστ έχει τώρα το λόγο για την ΚΟΕ. Δεν περίμενα να μου φωνάξετε τόσο γρήγορα. Κοιτάξτε, εμένα όλο αυτό το θέμα της ασφάλειας του διαδικτύου με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Κυρίως διότι τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία χρόνια μάλιστα, έχουν προκύψει απειλές από ε, παρακολουθήσεις τηλεφωνημάτων, από αυτές ε, τις παρακολουθήσεις από τις ΗΠΑ. Έτσι λοιπόν η προστασία των ε, δεδομένων θεωρώ ότι δεν είναι εξασφαλισμένη. Βρίσκω λοιπόν ότι ο φορέας Ενίζα έχει πολύ σημαντικά καθήκοντα. Είναι λιγάκι σαν τον Δαβίδ που έχει να αντιμετωπίσει το Γολιάτ. Και γι' αυτό θέλω να ερωτήσω αυτό το θέμα της ασφάλειας του διαδικτύου. Πώς ακριβώς το αντιμετωπίζετε, όπως επίσης ε, γενικότερα την ε, ασφάλεια των δεδομένων. Νιώθετε αρκετά ισχυροί για να αντιμετωπίσετε αυτές τις ε, νέες απειλές. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Το δεύτερο βέβαια έχει σχέση με το ε, πακέτο προστασίας δεδομένων που έχει κατατεθεί στο Συμβούλιο και όχι όλοι έχουν στρέψει τα βλέμματα εκεί, το τι ακριβώς ε, θα γίνει. Στον γενικό κανονισμό τίθεται το ερώτημα ε, τι θα προκύψει τελικά και κατά την άποψή σας ποια είναι τα πιο σημαντικά θέματα που πρέπει να σωθούν από την τριμερή συνάντηση τον τριμερή διάλογο. Οι διαπραγματεύσεις αυτές ε, του ε, τριμερού ε, διαλόγου θα είναι πολύ σκληρές. Εγώ είμαι μέλο τη Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, Πολιτικών Ελευθεριών και πραγματικά με ενδιαφέρει πάρα πολύ το τι έχετε να πείτε επ' αυτού. Εκ μέρους λοιπόν της, του, της πολιτικής ομάδας EFDD, ο κύριος Ταμπουράνο. Θέλω να κάνω μια ερώτηση που έχει σχέση με την προστασία τη ιδιωτική σφαίρας των ε, πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοιτάξτε, μερικοί εξημών εδώ είμαστε νέοι και θα θέλαμε να γνωρίζουμε ε, τι έγινε κατά το παρελθόν και τι πρόκειται να κάνει ο φορέας σας για θέματα παρακολουθήσεις ε, τηλεφωνημάτων στην περίπτωση NSA, αλλά και της GCAKQ μια περίπτωση που έχει σχέση με την Μεγάλη Βρετανία και όλα αυτά απέδισαν εις βάρος των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ε, παρατηρήσεις Ο κύριος Έλερ έχει το λόγο. Πρόεδρε, νομίζω ότι τα σημαντικότερα ερωτήματα ετέθησαν και εδώ επιτρέψτε μου εκ μέρους Επιτροπής Ήτρε να σας ευχαριστήσω και να πω ότι χαιρετίζουμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι θα παραμείνετε διευθυντής αυτού του φορέα. Και δεν το λέω ε, για να σας φιλοφρονήσω, αλλά διότι το κοινοβούλιο αυτό ε, αγωνίστηκε σκληρά για να ανεωθεί η θητεία του ΕΝΙΖΑ. Θελήσαμε να αυξήσουμε μάλιστα και τον προϋπολογισμό σας, το καταφέραμε και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί υπήρξαν μεγάλες προσπάθειες των κρατών μελών να περιορίσουν το φορέα, να περικόψουν τον ε, προϋπολογισμό και σε φύσεως θέματα. Ήταν λοιπόν μια μεγάλη επιτυχία της Επιτρόπου κυρίας Κρούς και του Κοινοβουλίου που κατόρθωσαν να ενισχύσουν το ρόλο του ΕΝΙΖΑ και να υπάρχει έστω κάποια επαρκής ε, χρηματοδότηση. Εδώ λοιπόν θέλω να υπογραμμίσω για άλλη μια φορά ότι αυτή η υποστήριξή μας ήταν από όλα τα κόμματα και γι' αυτό χαιρόμαστε πάρα πολύ που ήρθατε και εδώ σήμερα. Εμείς κατά τα επόμενα έτη θα παρακολουθούμε τη δουλειά του ΕΝΙΖΑ. Εμείς θα συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε την υποστήριξή μας, κυρίως στις συζητήσεις που θα ακολουθήσουν για τα κράτη-μέλη σχετικά με μια νομοθετική ρύθμιση. Ε, παρακαλώ να δείξετε κατανόηση γιατί δεν έχω να θέσω ερώτηση, αλλά θα ήθελα να έχω πει αυτά που είπα. Πρόεδρος, η κυρία Νιουάν Χάουζεν. Ευχαριστώ πρόεδρε και σας ευχαριστούμε και εσάς για την εισήγησή σας. Είπατε ότι η μόνη σταθερή αίρια στον κυβερνοχώρο είναι οι ταχύτατες αλλαγές. Συμφωνώ ε, απόλυτα μαζί σας ε, σε αυτή την εποχή και οι αλλαγές αλλάζουν πολύ γρήγορα και είπατε ότι κατά τα επόμενα πέντε χρόνια ο φορέας σας ε, προτίθεται να αντιμετωπίσει τις ε, προκλήσεις, ε, να προσφέρει νέα γνώση και νέες λύσεις. Αυτό δείχνει μεγάλη αυτοπεποίθηση και θέλω να σας ρωτήσω, θαυμάζω βέβαια την αισιοδοξία σας, αλλά από πού την αντλείτε, γιατί άλλοι ομιλητές είπαν ήδη ότι υπάρχουν πάρα πολλοί εγκληματίες που περιφέρονται. Και βλέπω επίσης ότι θέλετε να στηρίξετε την στρατηγική iClouding, να προσφέρετε ε, τα απαραίτητα πρότυπα ασφαλείας. Βεβαίως όλα αυτά μπορούν να γίνουν αν υπάρξει συμμόρφωση των ε, ενδιαφερομένων. Θα υπάρξει αυτή και αν όχι, αν οι hacker δεν συμμορφωθούν, εσείς τι προτίθετε να κάνετε, γιατί φαντάζομαι ότι οι hacker δεν είναι από αυτούς που πρόκειται να συμμορφωθούν. Θα έχετε στη διάθεσή σας μόνο τη Europol ή έχετε και άλλες πηγές πληροφόρησης. Άλλος, παρακαλώ, επιθυμεί κάποιος άλλος να λάβει το λόγο από τα μέλη, δεν βλέπω. Άρα δηλαδή έχετε το λόγο να απαντήσετε κύριε Διευθυντά. Ευχαριστώ Πρόεδρε και επίσης ε, ευχαριστώ πολύ και για τις ερωτήσεις που ετέθησαν. Επιτρέψτε μου επίσης να σας ευχαριστήσω και για την υποστήριξη που μου προσφέρατε κατά τα τελευταία έτη, γιατί όπως είπε και ο κύριος ε, Έλα χρειάστηκε αρκετός καιρός ε, για να πάρουμε την ανανέωση της θητείας μας. Ε, νομίζω λοιπόν και ελπίζω ότι ε, θα μας στηρίξετε και όταν θα τεθεί το θέμα της ανανέωσης της θητείας μας μετά από κάποια χρόνια. Θα αναφερθώ τώρα στις ερωτήσεις. Ξεκινάω ε, με αυτήν που αφορούσε την οδηγία. Θα πω κάτι γενικότερο. Κοιτάξτε, όταν, κάνεις αυτή, όταν κάνει κανείς αυτή τη δουλειά, τίθεται πάντα το ερώτημα τι μπορεί να αυτορυθμιστεί στον κλάδο και πότε πρέπει να παρεμβαίνουν οι κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια. Η εμπειρία μας είναι από την κυβερνητική σκοπιά και του φορέα ότι δεν γίνονται αρκετά στα κράτη-μέλη και μέσα στον ίδιο τον κλάδο. Έτσι λοιπόν αυτό που θέλω να φέρω είναι τρία θέματα που είναι πολύ σημαντικά. Το ένα, η κυβερνητική δομή στην Ευρώπη. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι είναι πολύ σημαντικό σε κάθε κράτος μέλος να υπάρχει μια δομή για τη διαχείριση των κρίσεων και για κλιμάκωσή της. Ε, τα τελευταία πέντε χρόνια κάναμε μεγάλη εμπειρία σε τεχνικό επίπεδο ε, έχουμε τις ασκήσεις μας που παραλαμβάνουμε κάθε δύο χρόνια. Ε, έχουμε μια κοινή επιχείρηση Ευρωπαϊκής Ένωσης ΗΠΑ. Σε τεχνικό λοιπόν επίπεδο έχουμε βελτιωθεί. Και έχουμε και άλλες δομές που αφορούν ε, στην αντίδρασή μας. Αλλά η ερώτηση που ετέθη είναι τι θα γίνει σε περίπτωση κρίσης στην πληροφορική. Ε, και ποιον επίτροπο θα πάρει κανείς ε, μέσα στη νύχτα για να ε, τον βγάλει από το κρεβάτι του. Κοιτάξτε, αυτό, από αυτό δεν υπάρχει ακόμα απάντηση. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι για την αναφορά των ατυχημάτων. Αν θέλει κανείς και εσείς ως βουλευτές να πάρετε μια απόφαση χρειάζεστε δεδομένα και στατιστικές πληροφορίες. Αυτό που κάνουμε τώρα στο 13α άρθρο της ε, ανακοίνωσης της ε, τηλεπικοινωνιακής είναι ότι όταν υπάρχουν ατυχήματα υπάρχουν υπάροχοι του διαδικτύου και η δημοσίευση γίνεται ε, για περιπτώσεις της προηγούμενης χρονιάς. Βεβαίως το θέμα είναι τι γνωρίζουμε για τυχήματα στην κριτική μας υποδομή. Στον τραπεζικό τομέα, στον χρηματοψηφικό τομέα υπάρχουν ρυθμίσεις. Γενικά όμως δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες. Άρα δηλαδή τι το ερώτημα, τι είδους πληροφορίες χρειαζόμαστε και ποια τυχήματα θα πρέπει να αναφέρονται. Το δεύτερο λοιπόν θέμα είναι η αναφορά τυχημάτων. Και το τρίτο είναι η ανταλλαγή πληροφοριών. Η ανταλλαγή πληροφοριών ας πούμε ε, βασίζεται αυτή στην εμπιστοσύνη, άρα δηλαδή υπάρχει διαφορετικό επίπεδο ε, ε, διαδικτυακής ασφάλειας στα διάφορα κράτη-μέλη. Έχουμε διάφορα επίπεδα ανταλλαγής πληροφοριών και όταν πρόκειται για απόρριτες πληροφορίες διαβαθμισμένες, τότε αυτές προφανώς περιορίζονται σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Εδώ λοιπόν η μεγαλύτερη πρόκληση είναι ε, να έχουμε εμπιστοσύνη και από την άλλη αυτή κατά κάποιον τρόπο να μετατρέπεται σε νομοθεσία. Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι που μας αφορά. Έγινε επίσης ε, αναφορά στον κανονισμό προστασίας δεδομένων. Και να πω κάτι έτσι γενικότερο εδώ. Μία από τις βασικές μας αξίες είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων στην Ευρώπη. Και έχουμε βρει την κατάλληλη τεχνολογία που είναι παραδείγματος χάρη κωδικοποίηση ή ηλεκτρονικές ταυτότητες. Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε και αυτή υπάρχει για δέκα περίπου χρόνια είναι ότι βασικά δεν είμαστε σε θέση αυτές τις τεχνολογίες να τις ε, ε, μεταφράσουμε στην πραγματική μας ζωή. Ας πούμε η ηλεκτρονική υπογραφή δεν χρησιμοποιείται σε καθημερινή βάση. Αυτό λοιπόν που χρειαζόμαστε θα θυμάστε ότι πριν από κάποια χρόνια υπήρχε ένα σχετικό project, αλλά αυτό που συζητάμε επίσης Υπάρχουν λοιπόν ε, προβλήματα και για την ε, χρησιμοποίηση της κωδικοποίησης και της ε, ηλεκτρονικής υπογραφής στην καθημερινή μας ζωή. Κάτι άλλο, σχετικά με την ασφάλεια αναπερίπτωση θα δείτε πριν από 15 χρόνια δεν γινόταν καθόλου λόγος για την ασφάλεια των προϊόντων και υπήρξαν πολλές συζητήσεις για την ποιότητα του λογισμικού όπου είχαμε ένα μονοπάραχο ε, που πουλούσε ε, τα λογισμικά στην αγορά. Αν δείτε όμως ε, τον κλάδο του λογισμικού θα δείτε ότι εκεί έγιναν πάρα πολλές βελτιώσεις. Έχουμε πλέον κοινά κριτήρια τα οποία χρησιμοποιούνται σε πάρα πολλές περιπτώσεις, όχι βέβαια σε αρκετές και θέλουμε να βελτιωθεί η ασφάλεια. Σήμερα βέβαια ασφάλεια αφορά μόνο εκείνα τα προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται σε διαβαθμισμένες πληροφορίες κυβερνητικές. Αυτό δεν υπάρχει στην καθημερινότητα. Άρα δηλαδή στην αγορά κυκλοφορούν κάποια προϊόντα που δεν έχουν σχεδιαστεί όπως θα έπρεπε. Και αν δείτε λιγάκι ας πούμε τα κινητά σας, τα smartphones, δεν υπάρχει σε αυτά ασφάλεια. Είναι απλά ένας υπολογιστής που είναι φτηνός, με μικρή διάρκεια ζωής ε, και θέλουμε σε αυτό να υπάρξει ασφάλεια. Και εγώ λέω στους ενδιαφερόμενους να έρθουν να το συζητήσουμε. Υπάρχουν και κάποιες άλλες ερωτήσεις σχετικά με τις ε, ταχείες αλλαγές, τις βασικές ε, προκλήσεις. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχουμε πολλούς εμπειρογνώμονες και το πλεονέκτημά μας είναι ότι έχουμε υπαλλήλου από το δημόσιο τομέα, από τον κλάδο που είναι πραγματικά πολύ δυναμικοί, εμπειρογνώμονες λοιπόν που δουλεύουν στα προγράμματά μας με ιδιαίτερη τεχνογνωσία. Βασικά το πρόβλημα που έχουμε, άλλοι μιλάνε για προκλήσεις, είναι ο φιδωλός προϋπολογισμός. Αν δείτε τον αρχικό σχεδιασμό, δυστυχώς διαπραγματεύσει έλαβαν χώρα μεσούσεις της οικονομικής κρίσης. Καταλαβαίνω ότι τα κράτη-μέλη δεν έχουν πολλά χρήματα. Το θέμα είναι πώς ιεραρχεί κανείς τα προβλήματα. Οι δικές μας ε, οι προκλήσεις είναι ότι πρέπει να επιλέγουμε κάποια θέματα και κάνοντας αυτό αφήνουμε κάποια κατά μέρος. Πολλέ φορέ έχουμε ένα υπάλληλο που δουλεύει για ένα θέμα χωρί υποστήριξη γιατί δεν υπάρχουν χρήματα. Άρα δηλαδή είναι θέμα ιεράρχηση, μιλώντα για την εσωτερική αγορά και για την περίφημη πρωτοβουλία push and pull, σήμερα θα δείτε ότι χρησιμοποιούμε ό,τι μπορούμε στα διάφορα προϊόντα. Οτιδήποτε υπάρχουν προϊόντα τα οποία έχουν κανονικά σχεδιαστεί για τη μαζική αγορά. Αν δείτε τα επιχειρηματικά μοντέλα υπάρχουν κοινωνικά δίκτυα, εμπορικές ε, ανταλλαγές, ε, αναζήτηση. Υπάρχουν μεγάλοι παίκτες όπως η Amazon, το Facebook, η Microsoft, ε, η IBM, πολλοί. Το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε στην Ευρώπη αν δούμε λιγάκι τον κλάδο μας. Και το θετικό μήνυμα είναι ότι στην Ευρώπη έχουμε ε, πολύ καλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εταιρείε ε, που έχουν ε, και παλίλους από 20 μέχρι 50, δεν έχουμε όμως μεγάλους παίκτες. Δεν έχουμε λοιπόν συμβουλευτικό όργανο για, με εκπρόσωπο από τον κλάδο. Βεβαίως ε, υπάρχει για τους μεγάλους παίκτες, όχι όμως για τους μικρούς. Η διαδικασία είναι ότι παίρνουμε το input από τον κλάδο και από τον ακαδημαϊκό τομέα και έχουμε εκεί και τους καταναλωτές και αυτό το input το μεταφέρουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο και εκεί υπάρχουν εκπρόσωποι των κρατομελών και εκεί συζητάμε το πρόγραμμά μας εργασίας. Αυτό λοιπόν παίρνει τις επίκαιρες προκλήσεις, τις μετατρέπει σε συζήτηση και από αυτά τελικά καταλήγουμε στο δικό μας το πρόγραμμα εργασίας. Τώρα θα έρθω σε ένα άλλο θέμα το οποίο εντάσσεται μερικά μόνο στις δικές μας αρμοδιότητες. Αναφέρομαι ε, στην κατασκοπία και στην αποκαλούμενη υπόθεση Snowden της περσινής χρονιάς. Να σας εξηγήσω λιγάκι τις ε, προκλήσεις και τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα. Η πρόκληση στην κυβερνοασφάλεια είναι ότι για πρώτη φορά υπάρχει η ίδια τεχνολογία που, τις οποίες γίνεται χρήση και κατάχρηση σε όλους τους τομείς. Ενώ δηλαδή το εξής. Όταν μιλάμε για ηλεκτρονική τραπεζική, τότε μιλάμε και για κυβερνοέγκλημα. Όταν υπάρχει ένας ιός, αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλους τομείς. Αν θυμάστε, είχαμε ιούς το Stuxnet ε, που επιτέθηκε στο ποινικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά αυτό το ίδιο μπορεί να επιτεθεί και σε αστικές πολιτικές, πολιτικά συστήματα. Αν δείτε λιγάκι θέματα πολεμικά, εκεί γίνεται η χρήση της ίδιας πληροφορικής, των ίδιων πληροφορικών συστημάτων, άρα μπορεί να υπάρξει κατάχρηση. Το πρόβλημα είναι ότι η δική μας κοινωνία ε, συνεχίζει να υπάρχει με τον παραδοσιακό τρόπο. Έχουμε δίωξη του εγκλήματος, αστυνομία και κατόπιν υπάρχει και η πρόληψη. Αν δηλαδή τα βάλει κανείς παράλληλα, πρέπει κάτι να γίνει στην πρόληψη στον κυβερνοχώρο. Και μιλάμε λοιπόν για τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αντιδράσουμε. Αυτά όμως είναι εκτός των αρμοδιοτήτων του ΕΝΙΖΑ. Και μετά υπάρχει το ε, κυβερνοέγκλημα και κάπου αυτά δεν εντάσσονται στην κοινή αγορά και υπάρχουν άλλοι τομείς ε, όταν μιλάμε ας πούμε για κατασκοπία σε επίπεδο ΝΑΤΟ και ούτω καθεξής. Με λίγα λόγια, η δική μας αρμοδιότητα αφορά την πρόληψη. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να δούμε εμείς τι μπορούμε να κάνουμε για το έγκλημα, για την πρόληψη, για την προστασία των δεδομένων, κωδικοποίηση, ταυτότητες, όλα αυτά τα προληπτικά μέτρα μπορούμε να τα εφαρμόσουμε. Για το clouding τώρα. Το δικό μας το μοντέλο είναι το εξής. Με βάση την τεχνογνωσία που έχουμε συνεργαζόμαστε με τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Πού είναι εσείς, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι κυβερνήσεις, ο κλάδος και οι πολίτες. Δύσκολο βέβαια να έχουμε πρόσβαση στους ε, πολίτες. Εμείς στηρίζουμε τα κράτη-μέλη ε, θα τα στηρίξουμε τον Οκτώβριο. Εκεί α πούμε προβλέπεται μια πολύ μεγάλη εκδήλωση σε συνεργασία με τον κλάδο ε, και την κυβέρνηση εδώ των Βρυξελών. Και επειδή δεν μπορούμε να πλησιάσουμε τα 500 εκατομμύρια στην Ευρώπη, έχουμε τις ενώσεις και μέσα από αυτές δουλεύουμε. Ε, είχαμε και κάποιες επιτυχίες πέρσι, γιατί αν πλησιάσει κανείς ενώσει τα κράτη-μέλη, μπορεί να έχει ένα τρόπο συνδυτοποίησης, ευαισθητοποίησης και αυτό να μεταφέρει μέσα από τις ενώσεις. Όταν μιλάμε για το clouding, από το 9 μιλάμε με τον κλάδο, με ενώσεις του κλάδου, ας πούμε με την Ένωση Ασφάλειας του clouding. Ε, υπάρχουν και πολλές συμφωνίες για το πώς μπορεί να παρισφρήσει η ασφάλεια στο clouding και στα κοινωνικά δίκτυα. Ε, μία ιδέα είναι να υπάρχει πιστοποίηση. Και το ενδιαφέρον είναι ότι η πιστοποίηση και η έλεγχη ε, προσφέρονται από ιδιωτικές εταιρείες. Έτσι λοιπόν με το να φέρνει κανείς κοντά όλους αυτούς τους διαφορετικούς παίκτες μπορεί να πείσει τον κλάδο να χρησιμοποιεί αυτά τα συστήματα. Και εγώ οραματίζομαι να είμαστε ανταγωνιστικοί και με ασφάλεια. Αυτό το έχουμε στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας αλλά και της ε, πληροφορικής. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Διευθυντά. Ακούσατε από όλους μας ότι παράπονα δεν υπάρχουν, δεν εκφράστηκε κάποιο παράπονο, μόνο θετικές παρατηρήσεις ακούστηκαν. Και ήταν πάρα πολύ καλή η προσέγγισή σας, πλήρης, δώσατε αναλυτικές απαντήσεις, άρα είναι θετικό το αποτέλεσμα της συνάντησης αυτής, σας το λέω ειλικρινά. Σας ευχόμαστε λοιπόν κάθε επιτυχία για τη νέα σας θητεία. Κάθε επιτυχία, κύριε Διευθυντά, συγχαρητήρια. And uh, the last point for this Το τελευταίο για σήμερα, το πρωί, γιατί είναι πρωί ακόμα, είναι η οδηγία για τη διάδοση γεωσκοπικών δορυφορικών δεδομένων για εμπορικούς σκοπούς. Παρουσίαση από το Διευθυντή Φιλίπ Μπρουνέτ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλώς ήλθατε, κύριε Διευθυντά. Από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Επιχειρήσεις και Βιομηχανία της Ευρωπαϊκής επιτροπή. Η οδηγία αυτή μας ε, επιδόθηκε τον Ιούνιο με στόχο τη θέσπιση ενός ξεκάθαρου νομικού πλησίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για προϊόντα υψηλής ευκρίνειας, προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ευκρίνειας. Ο κύριος Νέλη Φερότσι, ο Επίτροπος για βιομηχανία και επιχειρήσεις θα τα ερωτήματά σας για το θέμα αυτό στη συνάντηση που θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα. Άρα θα μιλήσουμε και για την ανταγωνιστικότητα και για την επανεκβιομηχάνηση αλλά και για όλα τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη διάδοση των γεωσκοπικών δορυφορικών δεδομένων για εμπορικού σκοπού. Και όλα τα προβλήματα που έχουμε με το πρόγραμμα Galileo. Σας παρακαλώ λοιπόν να κάνετε την εναρκτήρια ομιλία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή Ήτρε για την πρόσκληση. Ήδη κατά το παρελθόν ε, λάβατε προτάσεις για τον Γκαλιό, το Κοπέρνικο, στα ερευνητικά προγράμματα σε θέματα διαστήματος. Φαντάζομαι λοιπόν ότι πολύ εύκολα θα εξοικειωθείτε και θα κατανοήσετε αυτή την πρόταση. Η διάδοση γεωσκοπικών δεδομένων, δεδομένων παρατήρησης της γης για εμπορικούς λόγους είναι ένας νέος πολύπλοκος τομέας, όμως πολλά υποσχόμενος ταυτόχρονα και από οικονομικής πλευράς και τεχνολογικής πλευράς. Είναι ένας πυλώνας των διαφορετικών δράσεων που αναλαμβάνουμε στο πλαίσιο των νέων διαστημικών πολιτικών σε επίπεδο κομισιών για την παρατήρηση της γης συγκεκριμένα και πρέπει να λάβετε υπόψη ότι οι τεχνικές αυτές είναι πρόκληση τεχνολογική και έντονη πολιτική απόχρωση έχουν, όμως το διάστημα, και αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα, πρέπει μέσω των εφαρμογών αυτών να είναι πιο κοντά ε, όσο γίνεται πιο κοντά στον πραγματικό κόσμο και να υπηρετεί τον πολίτη. Πολλά συστήματα και πολλές υπηρεσίες που πρόκειται από το διάστημα ε, είναι απαραίτητες σήμερα για την ε, ευημερία μας άμεσα ή έμεσα και ο διαστημικός τομέας επίσης είναι ένας μοχλός, σημαντικός μοχλός επιστημονικής προόδου μέσω της έρευνας με το οποίο συνδέεται, είναι και καταλήτης όμως για τη δημιουργία ανάντι θεμάτων και υπηρεσιών, ιδίω ε, με τη συνδρομή μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είναι ένα τομέα λοιπόν με πάρα πολύ μεγάλο αναπτυξιακό δυναμικό. Να δώσω ένα παράδειγμα της τηλεπικοινωνίες, την πλοήγηση, την παρατήρηση της γης. Οι υπηρεσίε, σε σχέση ακριβώ με το τελευταίο θέμα, είναι εργαλεία τα οποία είναι ήδη απαραίτητα Γνωρίζουμε για παράδειγμα τις μετρολογικές προβλέψεις, την παρακολούθηση περιβάλλοντος, τη διαχείριση κρίσεων, την παρακολούθηση φυσικών καταστροφών ή καταστροφών προκαλούμενων από τον άνθρωπο. Και θα αυξηθεί η σημασία στο μέλλον. Αυτό τι σημαίνει, ότι η ζήτηση για δεδομένα που είναι και η πρώτη ύλη αυτών των υπηρεσιών επίσης θα αυξηθεί. Εξού και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε έμφαση στην παρατήρηση της γης, τη γεωσκόπηση, με βάση κάποιες, κάποιους άξονες με τους οποίους προσεγγίζουμε το θέμα αυτό ως το δυνατόν πληρέστερα. Πρώτον, δρομολόγηση του προγράμματος Κοπέρνικος. Δεύτερον, συμβολή στη βιομηχανική πολιτική που έχει σημασία τα διαστημικά προγράμματα αλλά και για όλες τις εφαρμογές που απορρέουν από αυτά τα διαστημικά προγράμματα. Υπάρχει μάλιστα σχετική ανακοίνωση από το Φεβρουάριο του 2013 και τρίτο σημείο, προφανώς έρευνα. Χωρίς έρευνα δεν υπάρχει καινοτομία και πάντα μέσω της καινοτομίας ε, περνάει η κούρσα του διαστήματος και πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκή παρουσία στο διαστημικό τομέα. Για να αντιμετωπίσουμε επιτυχία της προκλήσεις ε, θέλουμε ε, να είναι ανταγωνιστική και εύρωστη, στέρεα αυτή η βιομηχανία. Και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να έχουμε και μια ευρωπαϊκή διαστημική πολιτική σε επίπεδο ένωσης η οποία θα είναι αξιόπιστη θα είναι προσαρμοσμένοι και ευθυγραμμισμένοι με αυτό που κάνουν άλλοι, όπως παραδείγματο οι Ηνωμένε Και βέβαια θα πρέπει επίσης να μπορεί να συμμετέχει στη γενική προσπάθεια και στους στόχους για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ήπειρό μα. Στόχος μας λοιπόν και οδηγία που θα σας παρουσιάσω ένα πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο, ένα περιβάλλον που μακροπρόθεσμα θα επιτρέπει η ευρωπαϊκή βιομηχανία, η ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία να αποκομίζει τα ίδια ωφέλη με την ανταγωνιστική διεθνή βιομηχανία και συγκεκριμένα κυρίως την αμερικανική. Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης που προανέφερα, ορίσαμε πέντε ειδικούς στόχους, μεταξύ των οποίων είναι η δημιουργία ενός ε, συνεπούς νομικού πλαισίου, ενός ρυθμιστικού πλαισίου που θα μπορούσε να αποτελέσει το σχεδιάγραμμα, το σχέδιο μιας ευρωπαϊκής ρυθμιστικής, διαστημικής ε, πολιτικής, τέλος πάντων ενός ευρωπαϊκού διαστημικού δικαίου. Αυτή η οδηγία την οποία θα σας παρουσιάσω πιο διεξοδικά σε λίγο είναι σημαντική διότι εντάσσεται στις πέντε αυτές δράσεις προτεραιότητας της ανακοίνωσης του Φεβρουαρίου. Πιστεύουμε ότι αν βελτιωθεί το ρυθμιστικό περιβάλλον, όλες οι επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη από το διάστημα και την ε, παροχή δεδομένων που παίρνονται από το διάστημα, είτε έμεσα είτε άμεσα, θα ωφεληθούν, θα αποφεληθούν από την κατάσταση όπου θα υπάρχει διαφάνεια, τα συστήματα και η προμή δεδομένων θα είναι εγγυημένοι και βιώσιμοι. Εύκολα καταλαβαίνει κανείς ότι δεν υπάρχει τίποτε χειρότερο από όταν κανείς είναι επιχειρηματίας να ε, συγκροτεί μια επιχείρηση η οποία παρέχει υπηρεσία που βασίζεται στην προμήθεια κάποιων δεδομένων και επειδή μονομερός ή μερικός έχει τροποποιηθεί ο κανονισμός, η ρύθμιση σε μια χώρα, να μην μπορεί να υπάρχει αυτή η προμήθεια των δεδομένων και έτσι η επένδυση να αποτυγχάνει και να μην παίρνει τα προϊόντα αυτά ο τελικός χρήστης. Αυτή η πρόταση οδηγίας είναι το πρώτο νομοθετικό σχέδιο το οποίο εκπονεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει να κάνει με τα οικονομικά παράγωγα του διαστήματος και που δεν αναφέρεται άμεσα στα δύο διαστημικά προγράμματα, τον Καλίλιο και τον Κοπέρνικος. Ούτε είναι τμήμα της ερευνητικής πολιτικής. στόχοι της οδηγίας, παραλαμβάνω, της είπα, τους είπα τους στόχους, είναι οι γενική στόχοι της βιομηχανικής διαστημικής πολιτικής, είναι πρόθεση της ανάπτυξης και των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη γεωσκόπηση ε, στις αγορές της Ευρώπης και ιδίως στην αγορά των υπηρεσιών, ώστε να ευνοηθεί η καινοτομία να έχουμε επιδόσεις ε, καλές σε αυτό τον τομέα, ώστε αυτές οι δραστηριότητες να αναπτυχθούν όχι μόνο στην ευρωπαϊκή αγορά, αλλά να μπορούν να εξαχθούν παράλληλα. Τέλος, η οδηγία πιστεύω ότι είναι και ένας από τους πυλώνες που θα πρέπει να ενισχύσει την μελλοντική ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό. Τι βλέπουμε λοιπόν σε παγκόσμιο επίπεδο. Η αγορά των ε, δεδομένων, των γεωσκοπικών, ε, αν αυξάνεται με ταχύτητα τους ρυθμούς ε, σε ολόκληρο τον πλανήτη. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις είναι μεγάλες, υπάρχουν όμως και πολλές που είναι πολύ μικρότερες σε μέγεθος. Ο ιστός των μικροεπιχειρήσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι άκρος εξαπλωμένος στον τομέα αυτό. Και είναι σε καλή θέση, αλλά πολύ πίσω σε σχέση με τις ΗΠΑ και αντιμετωπίζουμε μια μεγάλη αύξηση του ανταγωνισμού από τον Καναδά, από την Κίνα, αύριο από την Ινδία και, όπως είπα, και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με πάρα πολύ μεγάλη αύξηση μεγέθυνση του κλάδου αυτού. Επίσης, υπήρχε ένα σημείο που ήταν σημαντικό ότι τα κράτη-μέλη που διαθέτουν δυνατότητες δορυφορικών δεδομένων υψηλής ανάλυσης ε, η ευκρίνεια είναι λίγα. Τρία τον αριθμό. Αύριο πέντε. Τα κράτη-μέλη όμως όπου οι υπηρεσίες που βασίζονται σε αυτά τα δεδομένα που παρέχουν οι πέντε χώρες, οι, πάντων, οι φορείς εκμετάλλευσης πέντε χώρες, τα κράτη λοιπόν που ωφελούνται είναι 28, είναι όλα και τα 28 κράτη-μέλη της Ένωσης. Επομένως θα πρέπει να ε, μπορούν όλα αυτά τα δεδομένα να είναι ε, διαθέσιμα προς όλους. Έπρεπε λοιπόν να υπάρχει αυτή η ε, εγγυημένη κυκλοφορία των δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό, σε αυτό αποσκοπεί οδηγία. Με ποιο τρόπο. Πρώτον, με τη δημιουργία, με την καθιέρωση μάλλον ενός κοινού δεσμευτικού ορισμού για το τι εστί δορυφορικό δεδομένο υψηλής ανάλυσης. Βάση μετρήσιμων κριτήριων και δικτών που θα ισχύουν για όλα τα κράτη-μέλη. Μπορεί να σας φαίνεται αυτό προφανές. Μέχρι τώρα όμως ο ορισμός δεν υπήρχε. Οι ρυθμίσεις λοιπόν ε, για δεδομένα που εφαρμόζονται στην ίδια έννοια και δεν υπάρχει ίδιος ορισμός είναι αποτέλεσμα, ε, μάλλον έχει ως αποτέλεσμα κάποιες διαφορές και αυτό σίγουρα είναι επιζήμιο. Δεύτερος στόχος της οδηγίας, υποχρέωση να εξασφαλιστεί επαρκώς η διάδοση των δεδομένων αυτών όταν θα δετεθούν για πρώτη φορά ε, στο εμπόριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί στη συνέχεια η οδηγία θα ζητήσει. Άπαξ και έχουν επαληθευτεί τα δεδομένα αυτά και ένα κράτος μέλος ε, ε, τίθεται εγγυητής με βάση και τα κριτήρια της οδηγίας, τα υπόλοιπα κράτη-μέλη θα πρέπει να δεχθούν την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων των τρίτων, ίσως και σημαντικότερο, δεσμευτικοί κανόνες και πρότυπα διαφάνειας και ορατότητας ε, που θα πρέπει να εφαρμόζονται από τα κράτη-μέλη. Ήδη το ανέφερα το πρόβλημα αυτό. Πρέπει να υπάρχει προβλεψιμότητα. Όταν δηλαδή έχουμε μια εταιρεία ε, η οποία έχει συγκροτηθεί με βάση την πρώτη ύλη που είναι αυτά τα δεδομένα. Υπάρχει ένα είδος ασφάλειας εφοδιασμού που προεξοφλείται και είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε εκ των προτέρων ότι αυτά τα δεδομένα που εκμεταλλευόμαστε μπορούμε να τα έχουμε συνεχώς στη διάθεσή μας και στο μέλλον. Τελευταίο, και ολοκληρώνω με αυτό, αγαπητέ Πρόεδρε, επιλέξαμε την οδηγία ως μέσο, γιατί ξέρετε ότι υπάρχουν ε, τα κράτη που έχουν προμηθευτές γεωσκοπικών δορυφορικών δεδομένων, έχουν εφαρμόσει συστήματα ελέγχου των δεδομένων αυτών. Υπάρχουν κράτη-μέλη που θα κάνουν το ίδιο μελλοντικά, αλλά πολλά κράτη-μέλη δεν θα έχουν στη διάθεσή τους ε, αυτούς τους ε, προμηθευτές δεδομένων. Άρα ήταν σημαντικό να έχουμε μια οδηγία, γιατί ανάλογα με το βαθμό ανάπτυξη των ελέγχων στα κράτη-μέλη και τη παρουσία ή όχι προμηθευτών δεδομένων, τα κράτη-μέλη αυτά θα έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν τα στοιχεία τη οδηγία στο εθνικό δίκαιο. Αυτά τα οποία θεωρούν σκόπιμο να μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο. Εδώ ολοκληρώνω την παρουσίασή μου και είμαι βέβαια στη διάθεσή σας για να απαντήσω στι ερωτήσει σα. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Διευθυντά θα συζητήσουμε αυτά τα θέματα ευθύ αμέσω. Εκ μέρου του ΕΛΚ έχουμε την κυρία Αντζέλικα Νίμπλερ που ήταν και πρόεδρος της Επιτροπής μας πριν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν ένα θερμό ευχαριστώ για την ε, ενδελεχή ανάλυση σας, κυρίως όσον αφορά τα στοιχεία τα γεωσκοπικά. Τον Ιούνιο ε, συμμετείχα σε μία συνδιάσκεψη στο Μόναχο και εκεί είχαμε και πολλούς εκπροσώπους από μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα δεδομένα, τα κατέργαστα δεδομένα και πώς μπορεί κανείς να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτά. Θέλω να σας κάνω δύο ερωτήσεις. Μήπως μπορείτε να μας πείτε με ακρίβεια ποιες είναι τώρα οι μεγαλύτερες προκλήσεις έτσι ώστε από αυτά τα ακατέργαστα δεδομένα ε, να μπορεί κανείς να προσφέρει αυτές τις οικονομικές υπηρεσίες. Ε, είπατε ότι πρέπει να υπάρχει ένα γενικό πλαίσιο. Επιτόπου υπάρχουν ε, κάποια κέντρα ελέγχου. Σε εμάς το Μόναχο υπάρχει το πρόγραμμα Γαλιλαίος και το Κοπέρνικος. Αλλά το ερώτημα που τίθεται είναι σε τελική ανάλυση και όσον αφορά τον έλεγχο των ε, δεδομένων, ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση. Εσείς είπατε ότι οι επιχειρήσεις ε, πρέπει να προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες για τα ακατέργαστα δεδομένα, να υπάρχει μια εξασφάλιση συνεχούς ροής δεδομένων. Και θέλω να ρωτήσω ποιος θεσμός είναι κατ' ουσίαν αρμόδιος. Είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι η ΕΝΙΖΑ ή μήπως θα υπάρξουν νέοι θεσμοί από πλευράς ε, διαδικασίας. Ε, τι ακριβώς ε, γίνεται ανεξάρτητα από την τεχνολογία. Και το δεύτερο ερώτημα είναι τελικά όλα αυτά τα οποία μπορούμε να διαθέσουμε ως ακατέργαστα δεδομένα, πώς ε, τα παρουσιάζετε, πώς τα διατίθετε εσείς. Είπατε ότι υπάρχουν οι δορυφόροι, <clears throat> αλλά είμαστε 28 κράτη-μέλη. Και θέλω να ρωτήσω πώς μπορείτε να διασφαλίσετε ότι τα κράτη-μέλη όπου δεν υπάρχει ακόμα η βάση για την παροχή υπηρεσιών, να προκύψει αυτή η βάση στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης κοινή αγοράς. Αυτές είναι οι δύο ερωτήσεις μου. Ευχαριστούμε πολύ. Πατενόφσκι τώρα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τον ε, Διευθυντή για τη λεπτομερή περιγραφή που μας έκανε της οδηγίας που ετοιμάζεται αυτή την εποχή. Πράγματι είναι πολύ καλό να μπορούμε να έχουμε συγκεκριμένες περιγραφές, συγκεκριμένους ορισμούς για, τον, για την οδηγία, για το σκοπό της οδηγίας. Για τα γεωσκοπικά δεδομένα είναι πράγματι πολύ σημαντικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη δεν είναι οι μόνοι που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα. Είναι πολύ ευαίσθητα τα δεδομένα αυτά και γι' αυτό λέω ότι η διαχείρισή τους θα πρέπει να γίνεται βάσει συγκεκριμένων αρχών και κανόνων. Από την άλλη πλευρά, ξέρουμε ότι κάποιες οδηγίες μπορεί επίσης να δημιουργούν και διοικητικά προβλήματα, διοικητικούς φραγμούς και εμπόδια που να περιορίζουν την πρόσβαση στα δεδομένα. Και εκτός από αυτά που είπε η κυρία Νίμπλερ, εγώ έχω να ρωτήσω τα δεδομένα αυτά πώς θα χρησιμοποιούνται. Ποιος, ποιο θεσμικό όργανο είναι αυτό το οποίο θα διαχειρίζεται αυτό το τομέα. Εγώ θα πρότεινα να χρησιμοποιήσουμε ένα από τα ρυθμιστικά όργανα και αυτό να αναλάβει και τη διαχείριση αυτή. Και αυτό το λέω προκειμένου να μην δημιουργηθούν εμπόδια για τα κράτη-μέλη και να βασιζόμαστε πάντα σε σαφείς και ξεκάθαρους ορισμούς. Τα διοικητικά εμπόδια πάντως είναι ο μεγαλύτερος φόβος μου. Διότι η οδηγία μπορεί να ανοίξει μια μεγάλη αγορά για το μέλλον. Καλό είναι λοιπόν να μπορούμε να ελέγχουμε τα δεδομένα. Ευχαριστούμε. Εκ μέρους της ΚΟΕ τώρα, παρακαλώ. λέει ο Ευχαριστώ. Θέλω να ρωτήσω κατά πόσο κατάλαβα καλά. Πρόκειται για δεδομένα τα οποία συγκεντρώνονται με δαπάνη από τον Ευρωπαίο Φορολογούμενο και αν κατάλαβα καλά διατίθεται δωρεάν σε όλους. Καλό αυτό. Ακόμα και σε μεγάλους, μεγάλες εταιρείες που μετά κερδίζουν ένα σωρό χρήματα από αυτά. Οπότε η ερώτησή μου είναι, είναι λογικός αυτός ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε όταν κάνουμε περικοπές στον προπολογισμό και δεν έχουμε κέρδη από αυτά. Οι μεγάλοι εμπορικοί συνασπισμοί θα είχαν κάνει το ίδιο αν συγκέντρωναν αυτοί τα δεδομένα, θα τα διέθεταν δωρεάν στο δημόσιο τομέα. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να χρεώνουμε κάπως τις μεγάλες εταιρείες οι οποίες κερδίζουν τόσα πολλά χρήματα από τα δεδομένα αυτά που έχουν πληρώσει οι Ευρωπαίοι πολίτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για την ερώτησή σας. Άλλος. Θέλει κανείς άλλο το λόγο. Παρατηρήσεις. Όχι. Ωραία. Εσείς τώρα κύριε Διευθυντά για να απαντήσετε. Και για να κάνετε και ό,τι άλλο σχόλια θέλετε. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Τις αναφέρατε πώς θα διασφαλίσουμε τη διαφάνεια στις διαδικασίες που σήμερα υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί θα δώσει απάντηση και στις δύο άλλες ερωτήσεις που ακούσαμε. Κοιτάξτε, σήμερα σε τρεις χώρες μέλη έχουμε διαδικασίες, οι οποίες όμως αποκλίνουν μεταξύ τους, βασίζονται σε διαφορετικά κριτήρια, ε, περνάνε από διαφορετικά βήματα και δεν υπάρχει προβλεψιμότητα γιατί υπάρχουν ελάχιστα αντικειμενικά στοιχεία στις διαδικασίες αυτές. Καταλαβαίνετε επίσης ότι η οδηγία έχει να κάνει με ένα πολύ ευαίσθητο τομέα. Πρέπει αφενός μεν να διασφαλίσουμε την ε, διάδοση όσο γίνεται περισσότερο δεδομένων υψηλής ανάλυσης για εμπορικούς σκοπούς γιατί μόνο για εμπορικού σκοπούς προβλέπεται η οδηγία αυτή, ενώ από πολύ καλά ότι τα δεδομένα υψηλή ανάλυσης συμπεριλαμβάνουν και στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με την ασφάλεια αλλά και με την άμυνα. Συνεπώς χρειαζόμαστε ένα σύστημα το οποίο να έχει μια καλή ισορροπία και να επιτρέπει όσο γίνεται ευρύτερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, επιτρέποντας όμως από την άλλη μεριά στα κράτη-μέλη να προστατεύονται και να προστατεύουν και την άμυνά τους. Συνεπώς η πρόταση αυτή οδηγία τι λέει. Λέει στα κράτη-μέλη. Εσείς θα πρέπει πρώτον στις χώρες σας πρέπει να δημιουργήσετε διαδικασίες και μία αρχή πολύ συγκεκριμένα Πρόεδρε, Μπορείτε να στήσετε από το συνάδελφο, λέει ο κύριος Φόξ, να μιλάει στο τηλέφωνο εκτός αιθούσης παρακαλώ και όχι εδώ γιατί ενοχλεί και δεν είναι και ευγενικό απέναντι στον ομιλητή μας, τον προσκεκλημένο μας. Συνεχίζει ο κύριος Μπρουνέ. Έλεγα λοιπόν ότι πρόκειται για μια ισορροπία που θέλουμε να πετύχουμε ανάμεσα στα δεδομένα που δεν είναι ευαίσθητα από πλευράς ασφάλειας και άμυνας, αυτά λοιπόν ευρύτατα να κυκλοφορούν, αλλά από την άλλη μεριά να ξέρουμε εκ των προτέρων ποια είναι αυτά τα οποία είναι ευαίσθητα και τα οποία χρειάζονται κάποια άδεια για να κυκλοφορήσουν. Αυτό θέλουμε. Όταν λοιπόν τα κράτη-μέλη θα έχουν ορίσει ποια είναι εκείνη η διοικητική αρχή η οποία είναι υπεύθυνη για την επαλήθευση των δεδομένων, πρέπει να έχουμε μία διαδικασία σε δύο στάδια. Πρώτον, να έχουμε μια τυπολογία των δεδομένων, κατά πόσο είναι ευαίσθητα ή όχι, βάσει κατηγοριών κριτηρίων και αν η απάντηση είναι ότι ναι είναι ευαίσθητα, τότε να υπάρχει διαδικασία άδεια ή να υπάρχει μια αρχή που με αντικειμενικά πάλι κριτήρια να αποφασίζει ποιο τμήμα των ευαίσθητων αυτών δεδομένων μπορεί να κυκλοφορήσει και ποιο άλλο δεν μπορεί να κυκλοφορήσει. Και έπειτα, εφόσον όλα αυτά θα έχουν γίνει στη χώρα όπου είναι κατεστημένος και ο πάροχος των δεδομένων αυτών, σκεφτήκαμε ότι θα ήταν καλό από κοινού οποιοδήποτε χρήση σε οποιαδήποτε χώρα μέλη να μπορεί να χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά άπαξ και μία χώρα έχει επιτρέψει την κυκλοφορία τους. Εντάξει, δεν είμαι νομικό εγώ, εγώ πώ το κατάλαβα το σύστημα, κατάλαβα ως εξής, να εφαρμόζουμε όχι σε δικαστήριο, αλλά σε μία διοικητική αρχή την ε, απόφαση για το κασίς της Διζών. Δηλαδή ότι όταν σε μία χώρα μέλη μπορούν ελεύθερα να κυκλοφορήσουν κάποια δεδομένα, μπορούν να κυκλοφορήσουν και στις υπόλοιπε. Είναι προφανές και το είπατε και εσείς κυρία Νίβλερ, ότι το πρόβλημα των δεδομένων που κυκλοφορούν ελεύθερα σε τρίτες χώρες μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Αλλά γι' αυτό δεν μπορεί να κάνει τίποτα η οδηγία, το πρόβλημα υπάρχει ήδη. Αν κάποια ευαίσθητα δεδομένα ε, έχουν ε, κάποια χώρα μέλη έχει επιτρέψει να κυκλοφορούν ελεύθερα, ε, η οδηγία τι μπορεί να κάνει. Η οδηγία το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να ρυθμίζει τη λειτουργία των δεδομένων άπαξ και αυτά έχουν ελευθερωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κυκλοφορήσει ελεύθερα μετά από άδεια κάποιου κράτους μέλους. Χρειάζεται λοιπόν ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια και την προσβασιμότητα. Και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε ανάλογα με τα διάφορα συστήματα και θα εκτιμηθεί και διαφορετικά θέλουμε να περιορίσουμε την οδηγία σε γενικά κριτήρια ώστε κάθε χώρα μέλη ανάλογα με το είδος δεδομένων που εξετάζει να μπορεί να έχει και κάποιο περιθώριο λιγμών. Για παράδειγμα, ανάλογα με αυτό που θέλετε να δείτε, υπάρχει ορισμός για το οπτικό φάσμα 2,5 μέτρα ή ορισμοί για τις υπέρυθρες, αν θέλετε να κοιτάξετε δικές εγκαταστάσεις, τέτοιου είδους κριτήρια θα λαμβάνονται υπόψη. Αλλά εμείς δεν το ξέρουμε και κανείς δεν ξέρει εξάλλου σε 10 χρόνια ή σε 5 τι θα μπορούμε να δούμε, τι θα είναι διαθέσιμο. Το θέμα τώρα των ε, δημοσίων δεδομένων και των ιδιωτικών δεδομένων. Αποφασίσαμε στο σύστημα Κοπέρνικους ελεύθερη πρόσβαση δεδομένων οι Αμερικανοί έκαναν ακριβώς το ίδιο με το σύστημα Landsat. Και για να είμαστε σωστοί, γιατί θελήσαμε το Κοπέρνικος να είναι ανοιχτό σύστημα, είναι για να μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί με το Landsat. Γιατί, γιατί αν προσφέρετε πάρα πολλά δεδομένα, ελέγχετε και τις υπηρεσίες οι οποίες δημιουργούνται και οι οποίες χρειάζονται τα δεδομένα αυτά. Οπότε σε πάρα πολλές περιπτώσεις θέλουμε τα δεδομένα Κοπέρνικους να είναι τα δεδομένα αναφοράς που θα χρησιμοποιούν οι αυτές και όχι τόσο το Landsat. Και οι είναι δωρεάν. Ε, εμπορικό τμήμα είναι τα δεδομένα υψηλής ανάλυσης, για τα οποία το, σύστημα Lancet ή το Copernicus δεν θα τα προσφέρει για τις περισσότερες εφαρμογές ανοιχτές στο κοινό και βιομηχανικές, τα δεδομένα που δίνονται από τον Κοπέρνικο και το Λάντσετ θα επαρκούν. Ενώ για κάποιες πολύ συγκεκριμένες εφαρμογές θα χρειάζεται να προσφεύγουμε σε δεδομένα υψηλής ανάλυσης. Και μόνο σε αυτό το τομέα θα ρυθμίσουμε. Και για να απαντήσω στην ερώτησή σας, τα περισσότερα συστήματα υψηλής ε, ανάλυσης είναι είτε στρατιωτικά είτε εθνικά και άρα δεν θα εμπίπτουν στην οδηγία αυτή, γιατί η οδηγία αυτή ασχολείται μόνο με δεδομένα για εμπορικούς σκοπούς. Και τα δεδομένα τα εμπορικά πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν ήδη πάρα πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν τα δικά τους δεδομένα. Αυτά θα ρυθμίσουμε. Σας ευχαριστούμε, κύριε Φιλιμπρουνέ. Σας ευχαριστούμε τις παρατηρήσεις σας και για την παρουσίαση της νέας σας οδηγίας. Όπως είπατε, είναι πολύ σημαντικό εμείς να δούμε την τρέχουσα κατάσταση, το ρυθμιστικό πλαίσιο, την έλλειψη εμπιστοσύνης, διαφάνεια, προβλεψιμότητα και βέβαια βασικός στόχος ή το βασικό καθήκον και στόχος της οδηγίας είναι η δημιουργία ενός διαφανούς και συνεπού νομικού πλαισίου για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν σαφές το μήνυμα, σας ευχαριστώ πολύ για τις εξηγήσεις που μας δώσατε και που ήσασταν εδώ σήμερα. Σας ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι. Ναι, ναι. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα συναντηθούμε μετά από τρεις ώρες. 12 έπρεπε να κλείναμε, άρα ακριβώς στην ώρα μας ολοκληρώνουμε. Στις 3 θα επαναλάβουμε τις εργασίες μας. Ευχαριστώ.